Well, good morning, and gentlemen. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε σιγά σιγά την ωραία μας συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα οι διερμηνείς ε, να σας ενημερώσουμε ότι βρισκόμαστε στην 17η ημέρα κινητοποιήσεων. Ε, χωρίς ε, κάποια συνεννόηση με τη διοίκηση. Οπότε η διερμηνία θα σταματήσει ακριβώς το προβλεπόμενο ωράριο. 12 και 30 ακριβώς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν να ξεκινήσουμε γέρος, λέει ο πρόεδρος. Καλώς ορίζω τα μέλη της Επιτροπής μας, τους καλεσμένους μας και το ακροτήριό μας. Μετά λοιπόν από το εργαστήριο το οποίο κάναμε συνεχίζουμε με μια ακρόαση με τίτλο «Διδάγματα από τα Paradise Papers» θα έχουμε δύο πάνελ. Το ένα θα μας πει αν ε, υπάρχουν κάποια παραθυράκια στη φορολογική νομοθεσία και αν πρέπει να αναλυφθεί περαιτέρω δράση. Ο κύριος Αχίμ πρόστο από η κυρία Γκάρ Σάιτ, δημοσιογράφος του η κυρία Λουσία Ρόσελ, ερευνήτρια στο έργο καταπολεμώντας την φορολογική απάτη και ενδυνάμωση των ρυθμιστικών αρχών. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Θα ήθελα να πω βεβαίως πως ε, αν δεν το ξέρετε έγιναν και άλλες αποκαλύψεις ε, γύρω από τον Παναμά. Ε, η δεύτερη ακρόαση θα ασχοληθεί με τις επιθετικές προλογικές πρακτικές. Δύο πολυεθνικές, η McDonald's και η Nike, ε, έχουν στείλει εκπροσώπους τους ε, στην Επιτροπή. Είχαμε καλέσει και την Apple, αλλά είπαν ότι κολλείονται γιατί υπάρχει μια υπόθεση στην οποία έχουν προσφύγει κατά της Κομισιόν ενώπιον του δικαστηρίου. Η αντιπροσωπεία μας θα συναντηθεί με την Επιτροπή αυτή αρχές Ιουλίου στις ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον. Επίσης, η Apple έχει δεσμευτεί ότι όταν ληφθεί απόφαση θα έρθει στην Επιτροπή μας. Η ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Κέρινγκ ε, δεν δέχτηκε την ε, πρόσκλησή μας γιατί ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν ε, ήταν διαθέσιμος. Είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις και δεν μπορούσαν να στείλουν κάποιον άλλον. Θα αποφασίσουμε τη Δευτέρα οι συντονιστές ποια συνέχεια θα δοθεί, δηλαδή εάν θα μπορέσουμε να προτείνουμε μια άλλη ημερομηνία στον Όμιλο Κέρινγκ. Οι ενδιάμεσες εταιρείες Appleby και Baker McKenzie επίσης έχουν προσκληθεί αλλά αρνήθηκαν λέγοντας ε, πως υπάρχει ζήτημα εμπιστευτικότητας ε, παρά τις διαβεβαιώσεις μου πως οι Επιτροπή δεν ενδιαφέρονται για συγκεκριμένους ε, πελάτες τους και ότι μπορούν βεβαίως πάντα να μην απαντήσουν εάν θεωρούν ότι αυτό πρέπει να κάνουν οι συντονιστές θα ζητήσουν τη συνέχεια θα δοθεί. Half Επίσης θεωρώ απαράδεκτο μια εταιρεία να μην ε, παρουσιάζεται σε μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι η διαφάνεια θα πρέπει να είναι κύρια αξία κάθε, αξία εταιρείας. Και εδώ πέρα θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Nike και της McDonald's. Με το να μην έρθουν στην ακρόαση η Applebee και η Baker McKenzie φαίνεται ότι δεν θεωρούν απαραίτητο να αντιδράσουν ε, στα δημοσιεύματα του τύπου για τα Paradise Papers. Βεβαίως η σιωπή αφήνει περιθώρια οποιασδήποτε ερμηνείας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα συζητηθούν οι εταιρείε αυτές από εμάς. Η ανταλλαγή απόψεων στο πρώτο πάνελ, ειδικά με μία δημοσιογράφο που είχε γράψει για αυτά τα θέματα, μπορεί επίσης να εστιάσει και σε αυτές. Είχαμε αποστείλει γραπτές ερωτήσεις, κάποιες απαντήσεις κρεμούν ακόμα. Οι γραπτέ απαντήσεις οι οποίες λάβαμε έχουν ήδη αποσταλεί σε όλους τους βουλευτές και θα είναι διαθέσιμες στο site της Επιτροπής μας μετά από την ακρόαση. Οπότε, να σας παρουσιάσω τώρα τους ομιλητές του πρώτου πάνελ, ο κύριος Αχίμ Προς. Διευθυντής του Τμήματος Διεθνούς Φορολογικής Συνεργασίας ε, στον ΩΣΑ και η κυρία Τζουλιέτ Γκάρσαϊντ, δημοσιογράφος ε, του Guardian για το θέμα αυτό και η κυρία Λουσία Ροσέλ Φλόρες ερευνητής ε, στο έργο καταπολέμηση της ε, φορολογικής απάτης και ενδυνάμωση των ρυθμιστικών αρχών. Θα έχουν λοιπόν λίγο χρόνο να απαντήσουν και μετά θα δεχτούν, να κάνουν μια αρχική τοποθέτηση και μετά θα δεχτούν ερωτήσει για να απαντήσουν. Κύριε Προς, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που δεν απάντησα γραπτό, Θα απαντήσω στα πέντε λεπτά που έχω. Οπότε, τέσσερα σημεία θα ήθελα να καλύψω. Το, η φορολογία των επιχειρήσεων που βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε. Δεύτερον, τα BEPS και αν υπάρχουν κάποιες σχετικές δομές, να δούμε πού βρισκόμαστε όσον αφορά τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Και τέλος, εάν ε, μου επιτρέπετε, τι μπορεί να γίνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο μετά τα Paradise Papers. Ξεκινώντας με κάποιους αριθμούς ε, και το τι σημαίνει η φορολογία επιχειρήσεων. Η φορολογία επιχειρήσεων μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Εάν δείτε τους αριθμούς, γεγονός είναι ότι το ύψος φορολογίας έχει πέσει πολύ στις χώρες του ΩΣΑ. Το 2000 είχαμε 32% και το 2018 βρισκόμαστε στο 23% κατά μέσο Αυτό κυρίως προ της ε, οικονομική κρίση όπου είχαμε μια σταθεροποίηση και τώρα έχουμε ξανά μια πτώση. Ε, αυτό το βλέπουμε ειδικά σε μεγάλες χώρες, σε Γαλλία, ΗΠΑ, οπότε δεν είναι μόνο οι μικρές οικονομίες που το κάνουν, είναι γενικό το φαινόμενο. Οπότε, εάν τα δείτε σήμερα, θα δείτε 22 χώρες του ΩΣΑ που έχουν ένα μέσο όρο εταιρικής φορολογίας στο 22% ή χαμηλότερα. Ταυτόχρονα το ποσοστό της ε, φορολογίας επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι σχετικά σταθερό. Και έχουμε αυτό το παράδοξο. Ως ποσοστό των εσόδων του κράτους έχει πέσει η φορολογία επιχειρήσεων, αλλά εξακολουθεί να είναι μεγάλο. Είναι 20% Οπότε οι χώρε εξακολουθούν να χρειάζονται τη φορολογία επιχειρήσεων και βεβαίω ε, την προηγούμενη εβδομάδα ε, μα ρώτησαν γιατί ανησυχούμε καν για το BEPS, ε, γιατί είναι σχετικά μικρά τα έσοδα και πρέπει να ανησυχούμε για κάτι άλλο εκτό από την φορολογία επιχειρήσεων. Αλλά είπαμε ότι γύρω στο 10% των, της φορολογίας των επιχειρήσεων κινδυνεύει, δηλαδή μιλάμε για, 200, για 240 δισεκατομμύρια παγκοσμίω. Οπότε είναι αρκετά μεγάλο το ποσό και ειδικά εκτό τη Ευρώπη πολλέ από τι αναψόμενε χώρε βασίζονται πολύ περισσότερο στην φορολογία των επιχειρήσεων. Οπότε αυτό πλήττει κυρίω τι αναπτυσσόμενε χώρε περισσότερο από τον ΩΣΑ. Αυτά λοιπόν για τα δεδομένα. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω που βρισκόμαστε με τα BEPS, αν έχουμε τελειώσει, αν χρειάζεται να κάνουμε κάτι περισσότερο. Εδώ, χωρίς να περάσουμε στα 15 σημεία δράσης, ε, τα, τις τέσσερις ελάχιστες προδιαγραφές κτλ. Το BEPS ακριβώς είχε στόχο να σταματήσει τον φορολογικό σχεδιασμό με βάση την έλλειψη διαφάνειας, την έλλειψη ουσίας και τρίτον τα παραθυράκια και την ασυνέπεια μεταξύ χωρών. Εδώ πέρα έχει γίνει τεράστια πρόοδο χωρίς να τα αναφέρω όλα. Λοιπόν, το θέμα δεν αφορά το ύψος ε, της ε, φορολογίας Οπότε αν τώρα θέλει κανείς να είναι σε ένα περιβάλλον χαμηλής φορολογίας, θα πρέπει να είναι εκεί και θα το ξέρουν όλοι, όλες οι φορολογικές αρχές. Είναι λοιπόν κάπως νωρίς να κρίνουμε γιατί η διαδικασία εφαρμογής συνεχίζεται και έχουμε τις πρώτες ε, εκθέσεις ε, αναχώρα οι οποίες ανταλλάσσονται μεταξύ των χωρών οπότε τώρα για πρώτη φορά λαμβάνουν τις ε, πληροφορίες οι χώρες, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Αλλά υπάρχουν κάποια ερωτήματα, ζητήσαμε αρκετή ουσία, πρέπει να σκεφτούμε το ύψος της φορολογίας. Υπάρχουν περιορισμοί στην Ευρώπη, παραδείγματο χάρη να, να μην είναι αποτελεσματικοί οι κανόνες, γιατί βεβαίως ε, υπάρχουν και κάποιες αποφάσεις που πρέπει να είναι συνεπείς με κάποιες ελευθερίες και βεβαίω πρέπει να δούμε και το κόστος της συμμόρφωσης και όλα αυτά ε, μακροπρόθεσμα. Εκεί είμαστε λοιπόν όσον αφορά τα BEPS ε, και αν μου επιτρέπετε δύο λόγια για τον ΩΣΑ και τις λίστες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς εστιάζουμε στην ε, διαφάνεια, έχουμε κάνει τα σχετικά. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ευρύτερη, δηλαδή ασχολούνται και με τα πράγματα τα οποία κάνουμε στα BEPS για τα οποία δεν έχουμε κατάλογο. Παραδείγματο χάρη, όταν εξετάζουμε τι φορολογικέ πρακτικέ, εμεί κοιτάμε όλε τι χώρε και δεν γίνεται διάκριση μεταξύ κρατών μελών και μη. Παραδείγματο χάρη, κοιτάμε και κοιτάμε ότι η Γαλλία έχει ένα λεγόμενο patent box το οποίο δεν συμφωνεί με του κανόνε Και βεβαίως ε, το ερώτημα είναι το τι μπορεί να γίνει ως αποτέλεσμα των Paradise Papers. Υπάρχουν ζητήματα διαφάνειας οπωσδήποτε. Υπάρχει η συζήτηση για τον, ε, τους πραγματικούς ε, ιδιοκτήτες. Υπάρχουν οι κανόνες υποχρεωτικής αποκάλυψης κάτι το οποίο υπήρχε στο Ηνωμένο Βασίλειο, τώρα υπάρχει στην Ευρώπη και ευρύτερα και βεβαίως το τι θα ισχύσει και ε, αλλού. Λοιπόν, αυτά θα σταματήσω εδώ για την ώρα. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η κυρία δημοσιογράφος. Ευχαριστώ που με καλέσατε να συμβάλλω στη συζήτηση και εγγράφαμε στον Guardian για τα Paradise και πριν για τα Panama και τώρα για το Δάφνη. Ε, οπότε τώρα συνεργαζόμαστε και συνεχίζουμε όλα αυτά ε, και για την καρουαναγκαλήσια και επίσης ε, προχωρούν παράλληλα αυτές οι τρεις έρευνες να σας πω για τις νομικές δυσκολίες που υπάρχουν για τους δημοσιογράφους όσον αφορά τέτοιε έρευνες και επίσης νομίζω ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις για μένα όσον αφορά αυτά τα οποία εμφανίζονται εδώ στα Panama Papers, τι γίνεται με την Applebee Ευχαρίστω λοιπόν να τα συζητήσουμε. Οπότε μου είπατε πως ε, αξιολογώ την προστασία των δημοσιογράφων όσον αφορά τη, ε, τις έρευνες που κάνουμε για τέτοιου είδους ε, φορολογικές στρατηγικές και οπότε θα πρέπει να ξεχνάμε τι γίνεται με τους δημοσιογράφους που έρευνουν τη διαφθορά. Υπάρχουν απειλές, υπάρχει παραπομπή στη δικαιοσύνη, μηνύσεις και είδατε γιατί έγινε και στη Μάλτα ακόμα χειρότερα και στον Guardian. Ποια είναι η εμπειρία μας υπάρχει ευθύνη να μπορούμε να ζητήσουμε απαντήσεις ε, εμεί που γράφουμε και πολλές φορές μας απειλούν με μηνύσεις πολύ συχνά και στη χώρα μας υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα τα οποία επιβάλλονται πριν την δημοσίευση αλλά επομένω υπάρχουν και τέτοιες νομικές απειλές και όταν έκανα κάποια σύγκριση με τη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, ε, δηλαδή σε τέτοιες συγκρίσεις μεταστάσεις τι γίνεται, είμαστε εμείς πιο ευάλωτοι. Να σας πω δύο παραδείγματα από τις απειλές που έχουμε στον Guardian. Είχαμε κάποια ξεχωρία εταιρεία, Applebee, θα την ξέρετε. Δεν έχουν έδρα στη χώρα μας, έχουν εγγραφεί στο Isle of Man και στις Βερμούδες και στην ίσο Τζέρσι. Και έγινε μια έρευνα από την Σιντότζε Τζάιντον, αλλά αποφάσισε η Appleby να συναντήσει τους δημοσιογράφους μας και του BBC στο Λονδίνο. Ζήτησαν αποζημίωση, μας ζήτησαν να τους δώσουμε τα Paradise Papers που είχαμε Επομένω, στο Κωσόβο υπήρχαν δύο ευρωπαϊκέ, εταιρείε, όλε οι άλλε εταιρείε ε, δεν αναμίχθηκαν σε αυτέ τι ε, απειλέ μηνύσεων από την Applebee. Και η Πρωθυπουργό είπε να τα δώσουμε, η Τερέζα Μέη, στο κοινοβούλιο. Είπε ότι θα πρέπει να δώσουμε τα χαρτιά στι διοκτικέ αρχέ. Όλα τα έγγραφα που είχαμε, καταλαβαίνετε αυτό ε, πόσο φοβίζει άλλους ε, πιθανούς ε, καταγγέλλοντες. Ναι, για τις φορολογικές αρχές γινόταν αυτό, αλλά ταυτόχρονα ήταν και εκφοβισμός προς τον Guardian. Να κόψουμε αυτές τις φορολογικές δημοσιογραφικές έρευνες, αυτό θα ωφελούσε και το κόμμα της Πρωθυπουργού και τις σχέσεις της ε, χώρας με τις ε, εταιρείε αυτές, τις ε, πρώην απικίες. Όλα αυτά τον Νοέμβριο δώσαμε σκληρή μάχη να προστατεύσουμε τα έγγραφα, τις πηγές μας και κυρίως το δικαίωμα να συνεχιστεί η δημοσιογραφική έρευνα. Τελικά συμβαστήκαμε με την Appleby και εμείς και το BBC για να προστατευτεί το δικαίωμα του δημοσιογράφου στην έρευνα. Και αν έρθουν σε μας κάποιοι με πληροφορίες, θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν κινδυνεύουν. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη για προστασία των πηγών μας και η η Guardian και το BBC γιατί ήταν στόχοι. Για δύο λόγους. Γιατί Είμαστε αγγλόφωνα έψιλον. Είμαστε οι πιο δυνατές φωνές στις καταγγελίες. Ε, έχουμε φήμη ότι είμαστε α, αντικειμενικοί, αλλά έχουμε πάρα πολύ αυστηρό δίκαιο που μας διέπει. δεν υπάρχει διάταξη αυτή για την ελευθερία του λόγου, το First Amendment, το αμερικανικό σε εμά, ούτε στην Γαλλία είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα. Οπότε, για να τώρα το δεύτερο παράδειγμα εκφοβισμού. Είναι πάρα πολύ ισχυρή και καλή οι δικηγόροι που ειδικεύονται στα τις συκοφαντίες και σε πάρα πολλές ε, χώρες τώρα έχουν κάποιους πλούσιους, Αζερμπατζάν, Κίνα και άλλα, που έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στέλνουν τα παιδιά τους εκεί στο σχολείο, επενδύουν και θέλουν να έχουν φορολογικά πλεονεκτήματα. Είναι πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει διάλογος αυτή πάνω κατευθείαν στους ε, δικηγόρους. Εντάξει, Είμαστε ισχυρή εφημερίδα. Αλλά δεν ισχύει αυτό για όλους. Δεν έχουν όλοι. Οι freelance, οι δημοσιογράφοι ας πούμε, δεν είναι τόσο ισχυροί. Και αυτό έχει επεκταθεί τώρα και εκτός Ευρώπης. Είδατε τι έγινε με την Καρουάνα Γκαλίτσια. Και επίσης έχουμε το φαινόμενο της χρυσή βίζα, και αυτά τα ερευνούσε η Δάφνη, αλλά απειλήθηκε με μήνυση για συκοφάντηση και στην Αγκόλα υπάρχει κάτι που μοιάζει με τα Paradise Paper για κάποιον Μάρκες και μιλούσαν για την λαιλάτιση του εθνικού πλούτου και τελικά ε, προσπάθησαν να καταφύγει σε διάφορες, διάφορα δικαστήρια ε, και του είπαν ότι αφού δεν κατοικεί στο Μένο Βασίλειο, γιατί προσφεύγει σε αγγλική δικηγορική εταιρεία. Επίσης, το συμπέρασμα είναι ότι δεν μπορεί μια αγγλική δικηγορική εταιρεία να απειλεί οποιονδήποτε με μήνυση στα βρετανικά δικαστήρια. Δεν μπορούν να διατυπώνουν απειλές για τα βρετανικά δικαστήρια. Τελικά ο νόμος προκαλεί εκφοβισμό, άρα πρέπει να τροποποιηθεί. Θα πρέπει αυτό να γίνει στην Ευρώπη. Σλαπ ονομάζεται αυτό στα αγγλικά όσον αφορά το δικαίωμα μήνυσης και υπάρχει, υπάρχουν αντίμετρα στη ΣΥΠΑ αλλά όχι στην Ευρώπη. Έχουμε πλησιάσει ευρωβουλευτές σχετικά με αυτό και θα μπορούσε αυτό το μέτρο να χρησιμοποιηθεί για να καταπολεμηθεί το ξέπλυμα χρήματο και οι φορολογικές απάτες. Δεν μπορώ παρά και πάλι να εκφράσω το θαυμασμό μου για τη δουλειά που κάνετε. Ανέκαθεν εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο σας στηρίζουμε στην προσπαθειά σας. Sorry. Uh, yeah, as said before, my name is Lucia I'm a political scientist. Καλημέρα σα. Ε, Λουσία Φλόρες ε, λέγομαι. Κάνω το διδακτορικό μου αυτήν την στιγμή ε, υπό την εποπτεία της κυρίας Ούγκερ, η οποία είναι υπεύθυνη για το ερευνητικό μας έργο. Εμείς εργαζόμαστε στην φοροαποφυγή, το ξέπλυμα χρήματος και η διαφορά μεταξύ των φύλων που προκύπτει από αυτό. Και εγώ ασχολούμαι κυρίως με την νομική και την πολιτική πτυχή. Θα ήθελα λοιπόν να σας αναφέρω πρώτα απ' όλα το τι ακριβώς είναι το έργο που το οποίο κάνουμε και το πώς μπορούν να μας βοηθήσουν τα Paradise Papers και γιατί χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Τα τελευταία 6 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βλέπει ανισότητες, ε, από πλευράς φίλου, γενεών, κινητικότητας ε, και ευκαιρίας. Ε, και ένας σημαντικός παράγων είναι η Το γεγονό ότι τα φορολογικά συστήματα φορολογούν περισσότερο την εργασία και την κατανάλωση από το κεφάλαιο. Και αυτό βεβαίω οφείλεται και στην φορολογική μυστικότητα. Σε συνδυασμό με την φορολογική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αντέδρασαν με καινοτομίε στον τομέα τη πολιτική, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ε, μιλάμε για μια μεγάλη αλλαγή στην φορολογική πολιτική. Είχαμε νέα έργα, νέα μέσα τα οποία ακριβώς τώρα αρχίζουν να εφαρμόζονται και το δικό μας ε, το ερευνητικό έργο μας δίνει ένα πλαίσιο για να αντιληφθούμε καλύτερα πώς έχουν τα πράγματα εξετάζοντας και τις ρυθμιστικές αρχές και τους ρυθμιζόμενους. Κοιτάμε δηλαδή τι αντίκτυπο έχουν οι νέοι κανόνες, ε, πώς ε, γίνεται η συστημική αλλαγή και παρέχουμε κάποιες δυνατότητες για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις. Σκοπεύουμε λοιπόν να δούμε το φορολογικό δίκαιο, την εξέλιξη της φορολογικής πολιτικής, φορολογικής διοίκησης και σκοπεύουμε να αξιολογήσουμε την χρησιμότητα και την δυνατότητα των εν μέσων να λύσουν προβλήματα. Θέλουμε, παραδείγματο χάρη, να αξιολογήσουμε την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, την αναφορά αναχώρα, το BEPS του ΟΣΑ και βεβαίω την ταυτοποίηση και αυτό θα γίνει με το να προσθέσουμε εμπειρικά στοιχεία σε μια πολλωμένη συζήτηση. Γι' αυτό όμως χρειάζομαστε περισσότερες πληροφορίες. Αντί να κοιτάμε προς τα πίσω, θέλουμε να αντιληφθούμε τα πλάθη του παρελθόντος και αυτό να αποτελέσει αφετηρία για το μέλλον. Και αυτό σημαίνει ανάλυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νομική προσαρμογή την προσαρμογή των φορολογουμένων, την προσαρμογή των ειδικών και της διοίκησης. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε καινοτόμε ε, προσεγγίσεις, κοινωνικο-οικονομικές ε, αναλύσεις, οικονομετρία. Αν μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο σιγά. Μα εγώ δεν σας καταλαβαίνω και είμαι ο ίδιος Άγγλος ε, με αυτά τα λαμπουρνέζικα που λέτε. Δεν έχουν καμία σχέση. Και δεν υπάρχει και πολιτική επιστήμη. Η πολιτική είναι τέχνη. Ναι, παρακαλώ να μιλάτε λίγο πιο ανθρώπινα. Ένας βασικός στόχος είναι να εξετάσουμε τα φορολογικά συστήματα ως οικοσυστήματα και να δούμε πως ε, οι επιχειρήσεις, οι ρυθμιστικές αρχές, οι λογιστές, οι δικηγόροι προσπαθούν να επιβιώσουν σε αυτό το νέο ρυθμιστικό καθεστώς και να βρουν ε, κάποια νέα σημεία επιβίωσης στην αγορά. Και ακριβώς θα μελετήσουμε τις αντιδράσεις ε, στην πολιτική και το τι αντίκτυπο έχει αυτό στο γενικότερο σύστημα. Θεωρούμε επίσης ότι τα νέα αριθμιστικά μέσα θα έχουν κάποια παραθυράκια τα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν. Όσον αφορά τα Paradise Papers, θεωρώ ότι μας δίνουν σημαντικά εμπειρικά στοιχεία γιατί βεβαίως οπωσδήποτε στα πανεπιστήμια και στην ε, έρευνα ήταν ένα θέμα η φορολογική παράδειση, αλλά βεβαίως θεωρία δεν υπάρχει χωρίς ε, στοιχεία. Δηλαδή υπήρχε πάντα το θέμα των ε, υπεράκτιων επενδύσεων, αλλά εδώ πέρα έχουμε μια αυξημένη διαφάνεια, έχει έρθει το θέμα στην δημοσιότητα και αποκαλύφθηκε ότι οι επενδύσεις αυτές δεν ήταν μόνο θέμα επιχειρήσεων, αλλά και ατόμων. Και αυτό έχει βεβαίως αυξήσει τον έλεγχο στον οποίο υποβάλλονται τα δημόσια πρόσωπα. Για εμάς λοιπόν τα Paradise Papers είναι σημαντικές πληροφορίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουμε την εμπειρική γνώση που θέλουμε να υπάρχει στη συζήτηση. Οι ερευνητές μας και άλλοι πανεπιστημιακοί έχουν πει ότι η διαφάνεια είναι ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθεί η φορολογική απάτη και τα Paradise Papers βεβαίως παρέχουν αυτή την απαραίτητη διαφάνεια. Αλλά αυτό δεν επαρκεί και για να καταπολεμηθεί η φορολογική απάτη χρειάζεται να υπάρξει ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της πολιτικές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση με τους ε, βουλευτές. Λοιπόν, ερώτηση ένα λεπτό ο καθένας. Ναι. Και μετά θα έχουμε τις απαντήσεις, αν επιτρέψει ο χρόνος, θα υπάρχει δυνατότητα να γίνουν και άλλες συμπληρωματικές ερωτήσεις, χωρίς να ξεπεραστεί ο συνολικός χρόνος. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, ο συνεισηγητής του ΕΛΚ, κ. Νίντερμαϊερ. Ευχαριστώ και εσάς που μιλήσατε τελευταίος και τελευταία μάλλον και όλα τα άλλα πρόσωπα. Έχουμε ρίξει το φως ιδιαίτερα στις μεγάλες εταιρείε και στο anti-money laundering και, στους, ε, και στις απάτες ΦΠΑ. Ε, Ένα θέμα δεν έχει καλυφθεί σε μεγάλη λεπτομέρεια. Ιδίως για υψηλού εισοδήματο ιδιώτες. Έχω λοιπόν τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, γνωρίζουμε ότι το πολιτικό και κοινωνικό κόστος των πολύ πλούσιων που μπορούν να καταφέρουν και πληρώνουν πάρα πολύ χαμηλές φορολογίες είναι βέβαια κάτι το οποίο οδηγεί σε φορολογική ανισότητα και έντονο ανικανοποιητό των υπολείπων. Σε ποιο βαθμό το θεωρείτε αυτό όχι μόνο κοινωνικό και πολιτικό θέμα, αλλά και, και ε, οικονομικό. Δεύτερο ερώτημα εδώ έχω το πρόβλημα της ατομικής φορολόγησης, αλλά και των εταιρικών δομών. Υπάρχουν νομοθετικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να σχεδιαστούν ειδικά για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, εάν συμφωνήσουμε ότι πρόκειται για κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και να αλλάξει. Και τέλος, ιδίω για τον ΟΣΑ η ερώτηση αυτή, πώς βλέπετε τη φορολογική στρατηγική των κυβερνήσεων απέναντι στο πρόβλημα των πλουσίων οι οποίοι είναι εισοδηματίες από μερίσματα και από κέρδη επιχειρήσεων και όχι από μισθούς και αμοιβέ. Για ένα λεπτό, μάλλον είναι πολλές οι ερωτήσεις. Α, τέσσερα λεπτά, τι ωραία. Έχω κάποιες σκέψεις. Πρώτα, υπάρχει ένα θέμα διαφάνειας πολύ σημαντικό θέμα. Αν εξετάσετε για παράδειγμα την περίπτωση των εγγράφων Παναμά, εάν το Common Reporting Standard, το κοινό πρότυπο δηλαδή για τις ε, ε, αναφορές είχε ισχύσει δεν θα υπήρχαν πολλά από αυτά τα πράγματα. Αυτόματο reporting δηλαδή για ε, τραπεζικούς λογαριασμούς. Ακόμα, τώρα που ισχύει ακόμα και ο Παναμά, ο Παναμάς αυτομάτως θα ανταλλάσσει πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς στον Παναμά μέσω ε, και για εισοδήματα από επιχειρήσεις που ε, είναι άλλοι οι κύριοι και οι δικαιούχοι των κερδών. Αυτά πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως, όχι μόνο ε, κατά γραμμά αλλά και κατά το πνεύμα. Και γι' αυτό εμείς, εμείς δηλαδή ο ΩΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε ε, θεσπίσει κανόνες αποκάλυψης, υποχρεωτικής αποκάλυψης, έτσι τα λέει ο ΩΣΑ, και αυτό είναι σημαντικό. Ε, μπορεί να γίνει περισσότερη δουλειά ακόμα, ώστε αυτοί που οφείλουν να γνωρίζουν και είναι πολλοί αποδέκτες αυτών των πληροφοριών, να γνωρίζουν όντως. Υπάρχει και το ζήτημα ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι Το ζήτημα ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι. Ε, το οποίο βέβαια πρέπει να ε, είναι και, να υπάρχει εκεί διαφάνεια. Δηλαδή να είναι γνωστή ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι. Πώ θα γίνει αυτό βεβαίω εάν υπάρχει, αν γίνεται τώρα στην ηλεκτρονική εποχή. Πρέπει να είναι στο διαδίκτυο και δεν μπορεί να είναι κρυμμένο κάπου. Εάν εξετάσετε και τα Paradise Papers, είναι και η φοροαποφυγή του ΦΠΑ. Και έχει δραστηριοποιηθεί τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί γίνεται προσπάθεια για να αυξηθεί η διαφάνεια. Βλέπουμε επίσης ως μια πολιτική αντίδραση, γιατί είναι πολύ δύσκολο τώρα πλέον να διακρίνει κανείς τον τόπο διαμονής από τον τροπεζικό λογαριασμό, Πολύ συχνά οι χώρες ανταγωνίζονται μεταξύ τους τώρα για να προσελκύσουν ε, ανθρώπους ε, για τόπο διαμονής. Πολλά μπορούν να γίνουν. Διότι συμφωνούμε όλοι δεν είναι μονάχα ζήτημα φορολογίας, είναι ζήτημα ισότητας, είναι ζήτημα εμπιστοσύνη ε, της κοινωνίας και γι' αυτό το φορολογικό, το φορολογικό ζήτημα είναι τόσο σημαντικό. Να μην εγκαταλείψουμε δηλαδή την διαφάνεια 100 χώρες συμμετέχουν τώρα. Πρέπει να συμμετέχουν, να συμμετέχουν όλες. Εάν το πρότυπο δεν αρκέσει, θα το ενισχύσουμε. Χρειαζόμαστε και την υποστήριξή σας. Και δεν είναι μόνο τομέας αυτός. Πρέπει να δούμε, να μην φτάσουμε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου θα προσπαθούμε όλοι να δίνουν φορολογικά κίνητρα σε κάποιες επιχειρήσεις και τελικώς όλοι να φορτώνουμε την φορολόγηση στην εργασία. Από τη στιγμή που έχει κανείς, που έχει φορολογική αρχή στα χέρια της πληροφορίες για όλα τα holding, από εκεί και πέρα είναι ζήτημα τη κυβέρνηση να αποφασίσει πόσο θα φορολογήσει την επιχείρηση, πόσο θα φορολογήσει το εισόδημα τη επιχείρηση, πόσο θα φορολογήσει την εργασία. Τώρα δημιουργούμε ένα σύστημα που θα δίνει τι πληροφορίε αυτέ, ότι τελικώ οι κυβερνήσει των χωρών να αποφασίζουν πώ μπορούν και τι θα φορολογήσουν. Ευχαριστώ. Πάνω από πέντε λεπτά πήρατε βέβαια. Ας προσπαθήσουμε να περιοριστούμε στις ερωτήσεις σε ένα λεπτό, σε συνολικά να μην περάσουμε τα πέντε λεπτά. Ορίστε. Ο κύριος Κόφουτ, ε, έχω διαβάσει την δήλωσή σας ε, γραπτή και γι' αυτό συγγνώμη, ε, ζητώ συγγνώμη και για την καθυστέρηση να προσέλθω. Για τα έγγραφα Paradise, ένα από τα σημεία που προκαλούν απογοήτευση είναι ότι κάποια από τα συστήματα αυτά φαίνεται να είναι εντός των πλαισίων τη νομιμότητα, αν και είναι βέβαια ανήθικα. Χρησιμοποιούν δηλαδή παραθυράκια του νόμου κλπ. Η πρώτη μου ερώτηση προς το πάνελ λοιπόν έχει ως εξή. Η υποβολή εκθέσεων αναχώρα θα είναι ένα πρότυπο διεθνώς για να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια φοροδιαφυγή. Πρώτη ερώτηση. Για την κυρία Γκάσάη τώρα έχω μια ερώτηση. Διάβασα και εγώ τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις που έχουμε υποβάλει. Αν σας ζητήσουμε να πείτε κάτι για την προστασία των καταγγελόντων, τι παραπάνω θα μπορούσατε να κάνετε εν ώψη και της εμπειρίας σας ως δημοσιογράφου. Δηλαδή η ερώτηση είναι μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι παραπάνω. Και τέλος, έχω διαβάσει και μια από τις ε, απαντήσεις σας που λέει, εκεί ρωτούμε δηλαδή για την οργάνωση Applebee που προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις όπως εξηγείται. Και μία από αυτές είναι η SCM Fides που ανήκει στην Aron Banks. Η τράπεζα που χρηματοδότησε το Brexit του κ. Κόπενς. Ποια είναι η διασύνδεση ανάμεσα σε αυτή την big business στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ε, υπηρεσίες και στον κόσμο των offshore. Θεωρείτε ότι είναι εφικτό να καλέσουμε ανθρώπους από τις επιχειρήσεις αυτές να καταθέσουν ε, μαρτυρίες ενώπιον της Επιτροπής για ζητήματα φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και τα άλλα ζητήματα που εξετάζουμε. Σας ευχαριστώ. Να αρχίσουμε την κυρία Ροσέλ. Όχι. Ο κύριος Πρόσ θα απαντήσω στο πρώτο τμήμα της ερώτησής σας. Το ερώτημα είναι, τα Paradise Papers έδειξαν κάποιες δομές φοροαποφυγής που φαίνεται, να, χωρίς να είναι ε, εγκληματικές ενέργειες, να οθούν τον νόμο στα όρια του. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν στη βάση της ε, υποβολής ε, εκθέσεων αναχώρα. Αυτές οι δομές δεν θα είναι πλέον δυνατόν να υπάρξουν ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε και ευρύτερα. Το reverse hybrid, για παράδειγμα, δεν θα υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστούν που έχουν εφαρμοστεί και έχουν απαγορευτεί τώρα και στις Ηνωμένες ε, Πολιτείες. Και οι διαρροές που έγιναν αναφέρονται σε προφορίες στο παρελθόν. Εάν προβάλλετε τώρα, κάνετε προβολή δηλαδή αυτών των πληροφοριών στο μέλλον, πολλέ από τι δομέ αυτέ δεν θα είναι δυνατέ πλέον. Δεύτερον, υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Πρώτα, η υποβολή εκθέσεων αναχώρα ανταλλάσσονται τώρα, τον Ιούνιο, για πρώτη φορά σε ολόκληρο τον κόσμο στην πράξη. Αν είστε λοιπόν μια εταιρεία όπως η Νίκε ή κάποια άλλη μεγάλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, στην Ινδία ή οπουδήποτε αλλού, η φορολογική αρχή όπου είστε εγκατεστημένος θα δει την έκθεση αναχώρα. Όλες δηλαδή οι φορολογικές αρχές, αν είναι 120 χώρες, είναι 120 φορολογικές αρχές που για πρώτη φορά βλέπουν τα πάντα. Όχι μόνο τι γίνεται στη δική τους χώρα, στη δική του επικράτεια, αλλά τι γίνεται και αλλού και τι γίνεται ενδιάμεσα και ποιο είναι το ποσοστό κέρδους που αποκτά τελικώ η εταιρεία. Αυτό θα είναι η τεράστια διαφορά. Και είναι ήδη τεράστια διαφορά. Πολλέ επιχειρήσει ήδη εγκαταλείπουν κάποιες ε, δομές, διότι δεν θέλουν να εξηγήσουν στις φορολογικές αρχές για ποιο λόγο έχουν όλες αυτές τις δομές σε διάφορες χώρες. Και στα υπόλοιπα, ας πούμε, 30 δευτερόλεπτα, το ζήτημα της δημοσίευση των εκθέσεων αναχώρα. Το έχουμε ήδη συζητήσει αυτό. Εμείς όσο όσα έχουμε κάποιες επιφυλάξει ό,τι αφορά την δημοσίευση, ε, την δημοσιοποίηση των ε, εκθέσεων αναχώρα. Τεχνικά θέματα, πολύ σύντομα τι μας ζήτησαν να κάνουμε όταν σχεδιάσαμε τις εκθέσεις αναχώρα. Μας ζήτησαν να φτιάξουμε κάτι για λογαριασμό των φορολογικών αρχών με master file κλπ. Και είπαμε εσείς χώρες να μην πηδήξετε να φτάσετε στα συμπεράσματα γιατί δεν ξέρετε ακόμη. Εάν τώρα τα δημοσιοποιήσετε όλα αυτά τότε καλείται το ίδιο το κοινό να αγνοήσει κάποια πράγματα και να καταλήξει ευθέως στα συμπεράσματα. Τώρα, υπάρχει και ένα δυναμικό διπλής φορολόγησης. μακρόν συζητήσαμε στον ΩΣΑ αν θα πρέπει να τα διαθέσουμε αυτά σε όλες τις χωρισμένες, γιατί πολλοί ανησυχούν για την διπλή φορολόγηση. Κάποια φορολογική αρχή μπορεί να κάνει κάποια φορολογική προσαρμογή όταν δεν υπάρχει, για παράδειγμα, ε, σύμβαση μη διπλή φορολόγηση με κάποια άλλη χώρα, μπορεί τελικώ να υποστεί διπλή φορολόγηση η επιχείρηση. Τέλο, υπάρχει ανησυχία εκτό Ευρώπη ότι όλοι, όλοι έχουμε κάνει κάποια συμφωνία. Αυτή είναι η συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, για την ώρα, το deal δηλαδή, που όμω δεν είναι δημόσιο κτήμα. Βεβαίω η Ευρώπη είναι απολύτω κυρίαρχη. Αν αποφασίσετε ε, να συνεχίσετε, να προχωρήσετε κι άλλο δηλαδή, αυτό είναι απόλυτο δικαίωμά σα. Αυτά είναι λίγα λόγια ω σκέψει από εμά, τον ΩΣΑ δηλαδή. Εσεί, κυρία Γκάσα, οι δημοσιογράφο, μίλησατε για του καταγγέλλοντε. Ε, προβλέπει η νομοθεσία για ειδική προστασία των καταγγελόντων η Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένω και νομική αρρωγή, δηλαδή πρόσφατα συνηγόρων. Είχα μια περίπτωση πρόσφατα όπου κάποιος ήλθε και με είδε και μου είπε με έχουν αναγκάσει να πάρω βαλίτσες με ρευστό σε ε, πτήσεις, σε αεροπλάνα για να πάω να λαδώσω ανθρώπους σε διάφορες χώρες. Τι θα γίνει αν με πιάσει η αστυνομία και θα χάσω τη δουλειά μου αν δεν το κάνω, μου είπα από την άλλη μεριά. Τους είπα λοιπόν στο πρόσωπο αυτό ότι εάν καταλήξεις στο δικαστήριο, οι δικηγόροι της Guardian δεν μπορούν να σε βοηθήσουν, θα πρέπει να πας να βρεις δικό σου συνήγορο. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολε αυτές οι ιστορίες που μαθαίνουμε να προβληθούν. Για να εξηγήσω τώρα πολύ σύντομα για τον Appleby, ε, που ε, ε, έκανε δηλαδή ήταν μια επιχείρηση θεματοφύλακα επιχειρήσεων, fiduciary business. Και είναι βέβαια αμφιλεγόμενο διότι είναι καλυμμένο από εμπιστευτικότητα. Ήταν θεματοφύλακας ε, επιχειρήσεων offshore και πρόσφερε εικονικούς διευθυντές για να καλύπτουν τους πραγματικούς διευθυντές και δικαιούχους. Η επιχειρήση γνώριζε Ποιοι ήταν οι ιδιοκτήτε, ενώ δεν γνώριζαν βεβαίω οι υπόλοιποι ούτε οι αρχέ ούτε το κοινό. Και αυτό που έγινε έκτοτε, αυτά είναι πριν από δύο χρόνια, αυτή η επιχείρηση επολύθη σε μια private equity και διαλύθηκε. Υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις τώρα που κάνουν τα ίδια σε ε, άλλες δικαιοδοσίες. Αγοράζουν άλλες φιντούρσεις, business και τις ενοποιούν με στόχο να αυξήσουν τα έσοδα. Τέτοιες επιχειρήσεις πάντως παίζουν πολύ ευαίσθητο ε, ρόλο και βρίσκονται υπό διαρκή πίεση να προσελκύσουν και άλλες πελάτες. Ελπίζω ότι η διαρεύνηση θα είναι πάρα πολύ ακριβή των ε, δραστηριοτήτων τους. Τέλος. Παρακαλώ προσπαθήστε να ολοκληρώσετε. Και η Aaron Banks έχει ε, μερίδιο στην Fidesz που κάνει fiduciary business και κάνει το ίδιο δηλαδή όπως η Φονσεκά στον Παναμά. Θα ήταν χρήσιμο να προσκαλέσετε κάποιον εκπρόσωπο αυτής της επιχείρησης. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σας παρακαλώ, ας παραμείνουμε στο ένα λεπτό, ιδίως για την υποβολή των ερωτήσεων και ιδίως αν έχετε παραπάνω από ε, μια ερωτήσεις. Εσείς τώρα, Μουρεσάν. Ευχαριστώ, σε όλες τις, ευχαριστώ όλες τις και τους ομιλητές, Στην κυρία Γκάρσαϊτ πρώτα, για το project Δάφνη που αναφέρατε προηγουμένως. Μπορείτε να μας πείτε κάποια από τα θέματα επί των οποίων εργάζεστε ε, ως συμμετέχουσα στο project Δάφνη με την έννοια της συνέχισης του έργου της Μαλτέζας δημοσιογράφου και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε. Θα ήθελα λοιπόν κάποιες ε, σχετικές πληροφορίε. Δεύτερον, είπατε ότι χρειαζόμαστε ε, νομοθεσία anti-slap στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσουμε δημοσιογράφους που διερευνούν φορολογικούς, ε, επιθετικούς μάλλον φορολογικούς σχεδιασμούς. Ποια άλλα νομοθετικά μέτρα θεωρείται αναγκαία για την προστασία των δημοσιογράφων όταν αυτοί διερευνούν τέτοια ευαίσθητα και ενδεχομένως επικίνδυνες τέτοιες και επικίνδυνες υποθέσεις. σε ό,τι αφορά την ρύθμιση. Κατ' επανάληψη μιλήσατε για την βιομηχανία offshore. Ποιες είναι οι νομικές δυσχέρειες που θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν οι αρχές και θα αντιμετωπίσουν οι Βρετανικές αρχές όταν δυστυχώς θα αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα πολλά θέματα θέσατε για το project Daphne. Η Μάλτα ενδιαφερόταν πολύ για κάποια μεγάλα θέματα και ιδίω ε, τις χρυσέ βίζες. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κάνει κάτι παρόμοιο, αλλά πολύ δικαίωμα διαμονής. Η Πορτογαλία πουλάει διαβατήρια και διαμονή. Η Αυστρία πουλάει διαμονή. Το ερώτημα είναι, ποιοι έλεγχοι έχουν γίνει για τους αγοραστές αυτών των ε, προξενικών θεωρήσεων, των χρυσών θεωρήσεων. Προέρχονται πολύ συχνά από τη Ρωσία, την πρώην Ένωση, από την Κίνα και ούτω καθεξής. Ξέρουμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, 3.000 οικογένειες ε, ε, έλαβαν το δικαίωμα να αγοράσουν έγκυο ιδιοκτησία μέχρι το 2015, χρησιμοποιώντας ε, χρήματα τα οποία η κυβέρνηση θεώρησε ότι είχαν ελέγξει την προέλευσή τους οι τράπεζες. και για πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, η κυβέρνηση θα πρέπει να γνωρίζει ποιοι έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό, ποιοι έρχονται ε, και εγκαθίστανται στην χώρα μέσα σε αυτό το σχήμα. Και θα πρέπει ε, να είναι γνωστά και τα ονόματά τους. Στη Μάλτα δημοσιεύονται τα ονόματα. Στην Κύπρο επίσης όσοι ζητούν ε, τέτοιες χρυσές θεωρήσεις. Υπάρχει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών που πρέπει να δημοσιευτεί. Το ίδιο στην Μάλτα φάνηκε η ανάγκη να συζητηθεί ένας οργανισμός, ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάποιο από την Τράπεζα τη Αγγλίας είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να αστυνομεύσουμε τι ίδιε τι τράπεζέ μα επαφιέμεθα στην ε, Αμερική στην ουσία να το κάνει, να κάνει τους ελέγχους αυτούς. Και η Μάλτα ως μια χώρα που δεν έχει ούτε την εμπειρία ούτε τους πόρους να καταπολεμήσει το ε, διεθνές ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Τα είδαμε αυτά, τι έγινε τελικώς σε βάρος της ε, δημοσιογράφου, της ε, Δάφνης. Και ούτω καθεξής. Το ε, ξέπλυμα χρήματος όμως είναι διαμεθοριακό θέμα, δεν γνωρίζει όρια, δεν γνωρίζει σύνορα και χρειαζόμαστε έναν ισχυρό οργανισμό διαμεθοριακού χαρακτήρα που να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Γιατί είναι δύσκολο οι εθνικέ αρχέ να αστυνομεύσουν την υπόθεση αυτή. Εξετάζουμε λοιπόν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο, εξετάζουμε τα χρυσά διαβατήρια, εξετάζουμε και οποιασδήποτε πολιτικέ επιρροέ στο έργο τη αστυνομία. Και ποιο εν τέλει στη Μάλτα μπορεί να έβαλε τη βόμβα. Τώρα για το ΣΛΑΠ δεν έχω να προτείνω κάποιο άλλο νομοθετικό μέτρο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η προστασία για, τη, για τους ανθρώπους που προσφέρουν πληροφορίες. Και, στη, και στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να φροντίσουμε να μην... Για, το, για τα υπερπόδια διαμερίσματα, πώς ήταν εκεί η ερώτησή σας. Οι συνέπειες ε, της Βρετανικής αποχώρησης του Brexit στις ε, Βρετανικές κτίσεις. βουλευτές από, την, ε, από τους συντηρητικούς αλλά και από αλλού ε, έχουν καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο για τις Βρετανικές κτήσεις μέχρι το 2021 και έχει περάσει το σχετικό νομοσχέδιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθεί να προβλέψει κάποιες προστασίες πριν να αποχωρήσουμε από την Ευρώπη, διότι ο κίνδυνος είναι ότι θα παραμείνουμε πολύ τρωτοί στο ε, ξέβλημα του δημόσιου χρήματος. και χρειάζεται ένα ε, ε, ισχυρός προμαχώνας απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο. Και τα σχετικά στοιχεία να είναι επιγραμμικά και προσβάσιμα. Έχετε να προσθέσετε κάτι, κύριε εκπρόσωπε του ΩΣΑ. Για τα διαβατήρια και τα πιστοποιητικά διαμονής έχουμε δει κάποια προγράμματα ανθρώπων που ζουν σε κάποια χώρα της Ευρώπης ε, να έχουν πιστοποιητικά διαμονής από άλλη ε, χώρα και τελικώς τα σχετικά έγγραφα να υποβάλλονται στη φορολογική αρχή άλλης χώρας. Αυτά τα στοιχεία τα συγκεντρώνουμε και θα προσπαθήσουμε να τα δημοσιεύσουμε. Τώρα για τους σοσιαλδημοκράτες, Ραμόν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα Ισπανικά θα διατυπώσω τις ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους. Για τον πρόσωπο του ΩΣΑ έχω τρεις ερωτήσεις. Σύντομες. Έχουμε την αίσθηση. Μετά τρία χρόνια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής ότι δεν προχωράμε και πολύ. Πρώτα πρώτα. Ρωτάω τον ΩΣΑ για να ξέρω αυτή η έκθεση αναχώρα πρόκειται να διευρυνθεί, να επεκταθεί. Τι εργαλεία, τι μέσα έχει ο ΖΑ, ούτω ώστε τελικά να το κάνουν περισσότερες εταιρείε. Άλλη ερώτηση. Πιστεύετε ότι πολιτικά θα έπρεπε τελικά τα πάμε καλά, έχουμε σωστή ρότα όσον αφορά το ποιε εταιρείε καλύπτονται. Είναι πολιτικά αποδοτικό αυτό για το μέλλον. Επίσης, αυτές οι γκρι, οι μαύρες λίστες, ωφελούν τέταρτον. Κυρία Γκάρσαϊτ, σε σχέση με την ε, αποκάλυψή σας, πολύ σημαντική. Εδώ στο Κοινοβουλίο πασχίζουμε για να υπάρξει μια οδηγία για προστασία των καταγγελόντων. Αυτό το οποίο είπατε, εγώ αυτό το κάνω τροπολογία. Σίγουρα θα το κάνω. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτούς που βοηθάνε το έγκλημα με ψευδές, κατά ψευδείς μηνύσεις. Κύριε Πρόσεχετε, εσείς πρώτος το λόγο. Α, από όσο κατάλαβα, έχω να σας απαντήσω τα εξής. Ναι, δεν έχουμε κάνει διαφορά στα τρία χρόνια. Θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ φόρο και εταιρικού φόρου. Άλλο το φυσικό πρόσωπο που κρύβει χρήματα σε κάποιο λογαριασμό εξωτερικό και τη εταιρεία που φόρο δεν λέω ότι θα πρέπει να αφήσουμε τον ένα ή τον άλλο. Θα πρέπει σαν τον γιατρό που εφαρμόζει άλλη αγωγή για κάθε ασθένεια να κάνουμε κι εμεί διαφοροποίηση. Οπότε, ε, όσον αφορά την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή με την ανταλλαγή πληροφοριών για του λογαριασμού, εκεί έχουμε κάνει πρόοδο. Κοιτάξτε τα νούμερα. Πολλέ χώρε έχουν μαζέψει 95 δι. Και αυτό γιατί ο κόσμος ξεσκεπάστηκε κατά κάποιο τρόπο. Έχει πληρώνει. Και όσον αφορά τι υπόλοιπε 50 χώρε που δεν το είχαν κάνει, θα το κάνουν το Σεπτέμβριο φέτο. Και οπότε έχουμε άλλε 100 χώρε που θα έχουν ανταλλαγή πληροφοριών για του λογαριασμού. Και με το Ενωμένο Βασίλειο και με άλλε χώρε. Οπότε, αν έχετε στον Παναμά, στην Ελβετία, όποιον έχετε λογαριασμό, οι σχετικέ πληροφορίε θα είναι αντικείμενο αυτή της ανταλλαγής προφορίας. Ένα, έχει γίνει η διαφορά. Φυσικά και πρέπει να γίνουν και άλλα. Όσον αφορά τώρα την έκθεση αναφορά, αναχώρα, δεν είναι εδώ το θέμα του ατομικού λογαριασμού. Αφορά μεγάλες πολυεθνικές. Όχι, δεν φοροδιαφεύγουν. Απλώς έχουν αυτές τις επιθετικές στρατηγικές, φορολογικές στρατηγικές. Έχουν ε, υποκαταστήματα, έχουν ε, θηγατρικές και πάνε εκεί που τι συμφέρει φορολογικά. Τι γίνεται τώρα, το είπαμε. Προσπαθούμε τώρα να καλύψουμε όλες τις εταιρείε που πρέπει να καλυφθούν. Και στο σύστημα τώρα έχουμε καλύψει 99% αυτών των εταιριών. ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία. 9% ναι, του ΑΕΠ καλύπτεται. Θέλουμε να επιταχύνουμε το ρυθμό της πρόοδος των ΩΣΑ, αλλά εν πρέπει όλα αυτά να ακολουθήσουν όλα τα βήματα από την ε, πρόταση μέχρι την νομοθέτηση και εφαρμογή. Αυτό έχουμε για το μέλλον ως πρόκληση. Τώρα, τι γίνεται με το κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε κάποιους ελάχιστους συντελεστές που να προβλέπονται. Αυτό σας απασχολεί και απασχολεί και εμάς. Όσον αφορά τους καταγγέλλοντες, ε, θα δώσω τη σκητάλη στην εκδεξιόν μου κυρία Γκάρσαϊτ. Ναι, ναι, ναι, σωστό να τους προστατεύουν τους καταγγέλλοντες παραπάνω και τους δημοσιογράφους παραπάνω όταν έχουν να κάνουν με απειλές μηνύσεων για σκοφατική δυσφήμιση. Και νομίζω ότι μέρος του προβλήματος είναι το εξής. Οι απειλές έρχονται από τους ζάπλουτους και κατευθύνονται κατά των δημοσιογράφων, ρεπόρτερ. Ευκολότερα βέβαια μπορεί να προστατευτεί ο Guardian παρά αυτοί που έχουν blog ή ε, ελεύθεροι επαγγελματίες δημοσιογράφοι πρέπει να βρουν τους δικούς τους δικηγόρους κλπ. Και πολλές φορές αυτοί ανακαλύπτουν τα Σκάνδα της διαφθοράς. Είδατε τι έγινε και με την ε, Μαλτέζα. Ε, δεν είχε και κανένα στρατό δικηγόρο να την προστατεύσει. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο πρόεδρος. Μάιτε. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Και εγώ να σας τα πω στα ισπανικά. Πρώτα-πρώτα, θαυμασμός και ευχαριστίες Προ την κυρία Γκρασάιτ και όλους τους του οποίου εκπροσωπεί. Είναι μια ομάδα βουλευτών, ευρωβουλευτών που ασχολούμεθα εντατικά, σοβαρά, εδώ και αρκετό χρόνο. Πρώτα-πρώτα, για να προχωρήσει αυτό το σχέδιο οδηγίας για προστασία των καταγγελόντων. Και τώρα προσπαθούμε συγκεκριμένα να δούμε το πώς θα παρακαμφθεί αυτό το βρώμικο παιχνίδι των ψευδομηνήσεων για να εμποδίσουν αυτούς τους ερευνητές να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι θέμα τελικά θωράξης της δημοκρατίας. Οπότε θα συνεχίσουμε σε αυτή την ερώτηση, σας διαβεβαιώνω. Πάντως, σε συνέχεια των όσων Χάρου, και έχω να πω τα εξή. Ξέρουμε ότι όσον αφορά την φοροδιαφυγή, γίνεται σε κάποιες χώρες που δεν είναι σε καμία μαύρη ή γκρι λίστα. Και έχουμε μια κάποια εκτίμηση του πόσοι είναι αυτοί που ξεπλένουν χρήματα και φοροδιαφεύγουν αυτό λόγω των Panama Papers, Paradise Papers κλπ. Οπότε, αν έχουμε μια ιδέα λοιπόν του πόσοι είναι αυτοί, είναι ακριβώς όπως τα είπε ο κύριος από τον ΩΣΑ. Για πετε μου. Όσον αφορά την αμοιβαία διοικητική συνδρομή, αρκεί δεν θα πρέπει να υπάρχει την υγεία του ΩΣΑ, ένα διεθνές όργανο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υποθεί ότι εμείς είμαστε ανυπόμονοι, απλώς ξέρουμε ότι θα πρέπει να σπεύσουμε δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο να αφορά την προσπάθειά μας για φόρο διαφυγή και ξέπλυμα. Πρόεδρος, ο επόμενος. Είναι ο κύριος Πρόσ. Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, συμφωνώ. 10%. 10% ε, χρησιμοποιούν από αυτό το φόρο. 240 δις ετησίως κάθε χρόνο. Η οικονομική μας ανάλυση αυτό υπέρνει ως βάση υπολογισμών. Πολλά λεφτά. Και τώρα έχουμε στοιχεία συνολικά αναχώρα. Και το 2019 θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για να δούμε αν έχουμε κάνει τη διαφορά με τις προσπάθειές μας. Είπαμε, επί τη βάση της εξολογησής μας, τα 240 ευρώ, τα οποία είναι απώλεια. Αυτοί που θα βρουν πληρώνουν και δεν πληρώνουν. Τόσο. Χρωστάνε. Αυτό θέλουμε να συρρυκνώσουμε, αυτό το ποσό. Και οι ε, εταιρείε μας λένε ότι το BEPS έκανε τη διαφορά. Τους άλλαξε τη συμπεριφορά και αυτοί που χαράσουν τις φορολογικές στρατηγικές το λαμβάνουν υπόψη. Τα ξέρουν οι φορολογικές αρχές. Και για πρώτη φορά θα είναι γνωστό το πού και τι γίνεται. Στα ισπανικά να σας απαντήσω, λέει κυρία Ροσέλ. Να σας πω δύο λόγια όσον αφορά το θέμα της, του υπολογισμού, της αξιολόγησης, το πόσα ξεπλένω και πόσο φοροδιαφεύγω. Δεν έχουμε ένα σίγουρο νούμερο, αλλά επεξεργαζόμαστε αυτά που τα λέμε μοντέλα κίνητρου με οικονομετρικά μοντέλα. Οπότε έχουμε κάποια προκαταρκτικά στοιχεία που μπορώ να σας τα στείλω. Τι εκτίμηση έχουμε κάνει για το ξέπλυμα και επίσης πόσα χρήματα φόρο διαφεύγουν. Αναχώρα και το σύνολο. Και έχουμε κάποια επιστημονικά μοντέλα, ούτως ώστε να το υπολογίσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η πράσινη μόλι Σκοτ Κέιτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους τα μέλη του πάνελ μας και ειδικά δημοσιογράφου του Guardian και θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του Brexit και της ε, φοροαποφυγής και τα κακά παιδιά του Brexit. Ξέρουμε ότι πολλοί από τους υπέρμαχους ε, του Brexit βρέθηκαν στα Paradise Papers και είχαν διάφορες υπεράκτιες εταιρείε. Βλέπουμε παραδείγματο χάρη ε, κάποιους ευρωβουλευτές, ο Τζέικο Μπρίσμοντ επίσης και αυτός βουλευτής ε, έχει εταιρείε στα Κέιμαν και τη Σιγκαπούρη. Ο Λόρδος Άσκροφτ έγινε γνωστός γιατί εκμεταλλεύτηκε το καθεστώς μη μόνιμου κατοίκου. Οπότε, Τζούλια, σας ερωτώ, αυτά τα κακά παιδιά του Brexit ε, έχουν σχέση με τα Paradise Papers. Θεωρείτε ότι ε, ο ρόλος τους σχετίζεται με αυτό και αυτό εννοούν όταν λένε να ανακτήσουμε τον έλεγχο. Μόλι να σε ευχαριστήσω και εγώ για την ε, δουλειά που έχει κάνει εδώ πέρα. Είσαι πολύ αποτελεσματική φωνή στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα ζητήματα ξεπλήματο χρήματο. Ναι, ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια σύνδεση. Αυτά είναι τα άτομα που εμφανίζονται συνεχώς όταν κοιτάμε το Ηνωμένο Βασίλειο και τα δεδομένα Οπότε μιλάμε για άτομα που συχνά ήταν και ταμείες του συντηρητικού κόμματος. Ο Λόρδος Φίνκ ε, ήταν στα πάνω ε, Papers. Ο Λόρδος Σόσκοφ επίσης στο Isle Ανεφέρατε τον κύριο Ρίσμογκ και αυτός το Isle έχει εταιρείε. Ο συνεταίρος του Jim Mellon επίσης ε, ε, ζει ε, στο Isle of Man για φορολογικούς λόγους. Οι αδερφοί Barclay, οι διοκτήτες της Telegraph που ήταν υπέρ του Brexit, επίσης βρέθηκαν στα Paradise Papers. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει μία σύνδεση. Το έχει πει ο Τζέρεμι Κόρμπιν ότι δηλαδή θέλουν το Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει ένας φορολογικός παράδεισος στα ανοιχτά της Ευρώπης. Ε, αυτή τη στιγμή σφίγγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Βρετανία θα γίνει πολύ πιο ευάλωτη σε τέτοιες ε, πιέσεις ε, ειδικά από αυτές τις επιθετικές ε, πρακτικές των ευγενών αυτών, των λόρδων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Και νομίζω καλό είναι να προσπαθήσουμε να προστατευτούμε και η διαφάνεια είναι νομίζω το μεγαλύτερο και επίσης και η δημοσίευση ε, όσων ε, έρχονται και αποκτούν άδεια διαμονής ε, λόγω επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει νομίζω μία σύνδεση άνθρωποι όπως ο Λόρδος Άσκροφ θεωρούν ότι το Brexit είναι μια ευκαιρία ε, για τις εταιρείε ε, με τις οποίες ε, βγάζουν τα λεφτά Να ρωτήσω κάτι επίσης για τις τράπεζες, γιατί και η χρηματοδότηση της εκστρατείας live.eu. Ο Άρον Banks mm. έχει μια εταιρεία χαρτοφυλακίου και εδώ και καιρό έχει μια εταιρεία επίσης ε, που λέγεται STM Feed, που αναλαμβάνει τέτοιες υπηρεσίες, δηλαδή να ιδρύει εταιρείε ε, υπεράκτιες για λογαριασμό των δικαιούχων για να κρύβουν την ταυτότητά τους. Οπότε αυτές οι εταιρείε ε, είναι ένας τρόπος να κρύβει κανείς το από πού έρχονται και πού πάνε τα λεφτά. Χρειάζεται λοιπόν νομίζω μια εξέταση αυτών των εταιριών και του τι συνέβη με την STM Fidex. Νομίζω πως ε, ο Observer ε, και η Κάρολ Κατουβόλιντα συγκεκριμένα ε, έχουν γράψει ενδιαφέροντα πράγματα τις τελευταίες εβδομάδες και βλέπουμε τώρα στοιχεία στενών δεσμών μεταξύ της ε, τράπεζας αυτής ε, της ε, ρωσικής πρεσβείας και νομίζω ότι το κοινοβούλιο μας και τα δύο κόμματα δεν θέλουν να ερευνήσουν τα θέματα αυτά για να βρεθούν στοιχεία συμπεγνία και δεν καταλαβαίνω γιατί εφόσον γίνεται στη ΣΥΠΑ, γιατί να μην γίνει και στην Βρετανία. Σας ευχαριστώ για την Γκουε Ματ Κάρθη. Ευχαριστώ και καλωσορίζω τους ομιλητές μας. Θα ήθελα να τους ρωτήσω για τις απόψεις τους για την διεθνή χρήση του μέσου της ε, Τη απόσβεσης ε, των άλλων ε, στοιχείων ε, ενεργητικού. Επίσης, ετέθη το ζήτημα της Apple και του συντελεστή φορολογίας που πληρώνει. Όπως είπατε, η Apple δεν ήρθε σήμερα, αλλά η μελέτη λέει πως ο συντελεστής φορολογίας Apple είναι γύρω στο 4% αλλά μπορεί τελικά να είναι και γύρω στο 1% και φαίνεται ότι τις ε, επιτρέπεται να, χρησιμο... να διαγράφει από τη φορολογική και 100% του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται ενδοετερικά για αγορά πνευματικής ιδιοκτησίας. Οπότε δεν πληρώνει τίποτα για τα κέρδη από τις πωλήσει. Τι πληρώνει τελικά το ίδιο ποσοστό φόρων που πλήρωνε και στο παρελθόν στην ε, Ιρλανδία. Και μας λένε στην Ιρλανδία ότι έχουν παρόμοιο φορολογικό καθεστώς με τις ΗΠΑ, την Βρετανία και αλλού. Αυτό το οποίο θέλουμε να ξέρουμε είναι οι δικές σας οι απόψεις για το εάν και κατά πόσον το φορολογικό καθεστώ της Ιρλανδίας ε, συγκρίνεται με την Βρετανία και ε, άλλες χώρες για το τι γίνεται με την πνευματική ιδιοκτησία. Σας ευχαριστώ. Ποιος θα απαντήσει αυτή την εύκολη ερώτηση. Ο κύριος από τον Όσα. Ε, δεν θα ήθελα, αλλά αφού δεν προσφέρεται κανείς άλλος. Δεν μπορώ να σχολιάσω, δεν ξέρω τα της Apple συγκεκριμένα, θα πρέπει να μιλήσετε με αυτούς. Ούτε την Ιρλανδική νομοθεσία καλύτερα από εσάς. κάτι το οποίο νομίζω θα έχει κάποια σχέση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΩΣΑ με τον κώδικα συμπεριφοράς και τις βλαπτικές πρακτικές κοιτάμε ακριβώς τη φορολογία της πνευματικής ιδιοκτησίας και αυτό το οποίο λέμε κατά κανόνα το κουτί γύρω από το κουτί το το κουτί το λεγόμενο με την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλαδή, εάν οι χώρες θέλουν να δώσουν κίνητρα στην έρευνα και την ανάπτυξη, κάτι το οποίο θέλουμε και οι περισσότερες χώρες το κάνουν και το κάνουν μέσω φορολογικών κινήτρων, όχι όλες, κάποιες, οι περισσότερες, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε τον παγκόσμιο χάρτη, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως ε, κατά κανόνα έχουμε ε, αυτή την χρήση. Τώρα, λοιπόν, ε, δεν λέμε ότι είναι επιβλαβές να φορολογείται χαμηλότερα η πνευματική ιδιοκτησία, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το όφελος που δίνεται είναι ανάλογο με την έρευνα και την ανάπτυξη. Δηλαδή, αν γίνεται και βεβαίω θα πρέπει να καθοριστεί πώ μεταφράζεται σε συντελεστή φορολογία, τότε η χώρα μπορεί να αποφασίσει τι συντελεστή θα εφαρμόσει. Θα ήταν επίμαχο αυτό και κάποιοι θα ήθελαν βεβαίως ε, να μην υπάρχουν ε, χαμηλότερε συντελεστέ για την πνευματική διοκτησία, αλλά εκεί πέρα κατέληξε η διεθνή κοινότητα στον ε ΠΕΠΣ. Το επανεξετάζουμε, κοιτάμε και το καθεστώ τη Ιρλανδία, το οποίο νομίζω συμμορφώνεται με τον ΩΣΑ, χωρί να ξέρω τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά είναι μια συνεχής πρόκληση από πλευρά ΩΣΑ αν δούμε δηλαδή από τη μία το θεμητό συμφέρον των χωρών να ενθαρρύνουν την έρευνα και ανάδειξη, αλλά να σταματήσουν ταυτόχρονα το φαινόμενο να μην ενθαρρύνουμε τελικά την έρευνα, αλλά να ενθαρρύνουμε τις ε, επιθετικές ε, φορολογικές πρακτικές. Αυτά χωρίς να ξέρω συγκεκριμένα τον ε, νόμο αυτόν. Σας ευχαριστώ. Κύριο Κόμπερν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τέτοια σοσιαλιστική μπουρδα δεν έχω ξανακούσει. Κύριε Σκότ Κέιτο, δεν είναι πολύ πατριωτικά αυτά τα οποία λέτε, αλλά δεν περίμενα και τίποτα διαφορετικό από εσάς. Αν ε, ψηφίζατε, βεβαίως ε, θα τα ξέρετε αυτά. Δεν είστε περήφανοι για την ε, Βρετανία και έχετε πρόβλημα με τον κύριο Μπάνξ, ο οποίος έδωσε λεφτά σε μια εκστρατεία γιατί πίστευε σε κάτι. Ο κύριος Σόρος, από ό,τι φαίνεται, στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς δεν κάνει ερωτήσεις για αυτόν. Ε, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτό, γιατί και αυτό στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διαφορέ τρέλες σας. Προσπαθεί να υπονομεύσει τη Βρετανική Δημοκρατία. Ναι, ναι, έρχομαι τώρα. Θα φτάσω και σε αυτό. Να επισημάνω ότι σύμφωνα με τον Βρετανικό νόμο, οι διευθυντές επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένοι να μειώσουν τους φόρους ε, στους μετόχους τους. Έτσι κάνουμε στη Βρετανία, γι' αυτό είναι επιτυχής η οικονομία μας. Τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας είναι ουσιαστική λειτουργία του κράτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι προστατεύει την ε, προστασία κάποιων δικαιωμάτων, όπως παραδείγματος χάρη τα, τα ζητήματα ιδιωτικότητας αλλά πάλι φόρου περνάει. Δεν σα ενδιαφέρει να προστατεύσετε την ιδιοκτησία. Το GDPR και ο φόρος ε, link είναι απλά ένας τρόπος να ε, μπείτε στα προσωπικά του καθενός. Και τι κάνετε, χρησιμοποιείτε τα Paradise Papers για πολιτικούς στόχους και από ό,τι ακούω δεν έχει γίνει κανένα δίκημα. Οπότε το ζήτημα εδώ πέρα είναι να μας πείτε τι ενάρετοι που είστε. Και θα ήθελα να ακούσω από την κυρία του Guardian πώς θεωρείτε ότι θα επιβιώσουν οι επιχειρήσεις εάν ο κάθε υπάλληλο αποκαλύπτει τα πάντα. Δηλαδή, για το όνομα του προφανώς δεν έχετε καμία εμπειρία από εταιρείε, αλλιώ θα συνειδητοποιήσετε ότι είναι αδύνατο να λειτουργήσει καμία επιχείρηση ή τράπεζα χωρίς εμπιστευτικότητα. Πρέπει να ε, συμμορφωθούν με τον νόμο. Δηλαδή, αν είναι να λένε τέτοια πράγματα, ε, πρέπει ακριβώς να αντιμετωπίζουν και τις συνέπειες του νόμου, όπως και οι δημοσιογράφοι. Έτσι, πρέπει να υπάρχουν συνέπειες, αλλιώς θα αρχίσετε την ε, δυσφήμιση χωρίς ε, καμία αναστολή. Ε, μα από πού να αρχίσω από όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ας δούμε το δικαίωμα να πληροφορούμε τον κόσμο για το τι γίνεται στις επιχειρήσεις και στις διάφορες δομές που ιδρύουν άτομα για να εξασφαλίσουν την περιουσία τους. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι δημόσιο κτήμα και πρέπει να προστατεύεται ο νόμο, από τον νόμο. Έχουμε δικαίωμα βέβαια ιδιωτικής σφαίρας, αλλά πρέπει να εξισορροπείται από το δημόσιο συμφέρον. Λέτε ότι δεν παρανόμησε κανείς στα Paradise Papers. Υπήρξαν περιπτώσεις φορό αποφυγής που θα μπορούσαν να αυθούν ενώπιον των δικαστηρίων και οι Βρετανικές φορολογικές αρχές εξετάζουν τα διάφορα συστήματα που ίσχυσαν εκεί στο Isle of Man με, ναι, για παράδειγμα, εκατοντάδες ε, ιδιωτικά αεροσκάφη τα οποία είναι καταχωρισμένα εκεί και δεν πληρώνουν ούτε μία λίρα φόρο. Είναι τόσο επιθετικός ο φορολογικός αυτός σχεδιασμός που ίσως και να έχουν υπερβεί τα όρια του νόμου. Ασφαλώς και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικές και προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την προσωπική σφαίρα των ανθρώπων και υπάρχουν μέτρα προστασίας τους είμαστε υποχρεωμένες να διαγράψουμε υλικό το οποίο ε, ε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει ενδιαφέρον για το κοινό, αλλά έχουμε και το καθήκον όταν μας υποβάλλονται πράγματα που ίσως με να, μην είναι παράνομα, αλλά σαφώς είναι αντίθετα με αυτά που θεωρεί η κοινωνία ότι θα πρέπει να γίνονται και ίσως ε, αυξάνουν την ανισότητα στην κοινωνία. Και όταν υπάρχουν συστήματα τα οποία ε, εξυπηρετούν τους πάρα πολύ πλούσιους και δεν μπορούν να τεθούν και στη διάθεση αυτών που δεν έχουν τη δυνατότητα να το πληρώσουν. Το ζήτημα δεν είναι μονάχα αν είναι παράνομη συμπεριφορά. Το ζήτημα είναι και αν υπάρχει ανήθικη, αντιδιοντολογική, επιθετική συμπεριφορά. Και εμείς ζητούμε να αλλάξει το σύστημα. Τα Paradise Papers έχουν δείξει ότι θα πρέπει να επιμένουμε να γίνουν μεταρρυθμίσεις και πολύ σωστά κάναμε Επανέρχεται ο κ. Κομπέρν. Ξεπερνούμε τα όρια του χρόνου. Γιατί δεν κυνηγάτε τον κύριο Σόρος. Γιατί δεν ρωτάτε... Ε, ο πρόεδρος Διακόπτη. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις ε, για τον κύριο Πρόσκη, και την κυρία Γκάρσαϊντ για τα αρχή αυτά, τα IBO. Τα πάντα papers βεβαίως αφορούσαν φορολογικούς ε, παραδείσου. Το μεγάλο όνομα από τις εταιρείε ήταν η Appleby και στον Παναμά η Mossack Fonseca. Η διάμεση, λοιπόν αυτοί ε, προσκλήθηκαν αλλά αρνήθηκαν από τις χθεσινές αποκαλύψεις φαίνεται πως ε, το ζήτημα αφορά ακριβώς ε, την αποκάλυψη των τελικών ε, δικαιούχων. Και θα πρέπει ακριβώς να υπάρχουν τέτοια μητρώα για να μπορούμε να βρούμε πολύ πιο εύκολα τους τελικούς δικαιούχους. Παραδείγματος χάρη έχουμε ε, ένα τέτοιο μητρό το οποίο θα τεθεί ενισχύ τον Ιούλιο του 2018 αλλά θα πρέπει να υπάρχει και δημόσια πρόσβαση σε αυτό το αρχείο για κάποιον ο οποίος έχει λόγο βεβαίως όπως παραδείγματος χάρη οι ερευνητές δημοσιογράφοι. Θεωρείτε ότι τα μητρώα αυτά προς τον ε, κύριο Πρόση ερώτηση επαρκούν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τα πραγματικών δικαιούχων. Και το ερώτημα είναι, θα μπορέσει όντω να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο αρχείο το πρόβλημα. Και το ερώτημα το οποίο έχω για την κυρία Γκάρσαϊντ είναι το εξή ακριβώς Αφορά την ε, δημόσια πρόσβαση στα μήτρο αυτά. Θα σας ε, βοηθήσει αυτό, θα αρκεί ή θα πρέπει να πάμε ακόμη παραπέρα θεωρείτε. Σας ευχαριστώ και ως προς. Ε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα εστιάσω στην φορολογική ε, σκοπιά γιατί οι συνάδελφοί μου δεν θα ήθελαν να επεκταθώ. Δύο παρατηρήσεις όχι μόνο λόγω των Paradise Papers αλλά και λόγω αυτών υπήρξε μια όθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΩΣΑ και καταλήξαμε σε αυτό το οποίο λέμε υποχρεωτική αποκάλυψη. Τώρα έχουν ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Εντάξει, βεβαίω πρέπει να εφαρμοστούν πρώτα, αλλά έχουν συμφωνηθεί ήδη. Και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιο ε, στην μία αδιαφανή offshore εταιρεία ως ενδιάμεσος, θα πρέπει να το αποκαλύψει αυτό στις αρχές της ε, χώρας σου και βεβαίως ε, στην χώρα στην οποία κατοικεί ο δικαιούχος. Αυτό είναι το ένα, είναι ευρωπαϊκό δίκαιο, μας έχει απασχολήσει και στον ΩΣΑ και πρέπει να καλύπτονται όλοι όσοι πρέπει να καλύπτονται από αυτά γιατί θα έχουμε κάποιες ε, καταστάσεις όπου οι άνθρωποι αυτοί δεν θα παραμείνουν στην Ευρώπη. Το ένα είναι αυτό το οποίο προωθούν οι G7, τα λοιπά. Και μετά για τους πραγματικούς δικαιούχους και το τι πρέπει να είναι διαθέσιμο. Ήδη έχουμε μια πρωτογραφή που απαιτεί να τηρούνται πληροφορίες ε, και για τους ιδιοκτήτες και για τα ε, λογιστικά αρχεία και να είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματο των φορολογικών αρχών. Ε, και αυτό σημαίνει σε 149 χώρε. Ουσιαστικά όλες οι χώρες που σας απασχολούν. Αυτό το εργαλείο είναι στη διάθεση των φορολογικών αρχών και τώρα εφαρμόζουμε την ε, προδιαγραφή του πραγματικού δικαιούχου και μπορείτε να δείτε αναχώρα ε, το πόσο προσπαθούμε να αποκτήσουμε τις πληροφορίες όχι μόνο για τον ε, νόμιμο αλλά και τον πραγματικό δικαιούχο και όπως σας είπα οι πληροφορίες αυτές δεν είναι σε ένα κομμάτι χαρτί αλλά ηλεκτρονικές, οπότε καλό είναι να είναι δομημένα τα δεδομένα. Για το αν θα πρέπει να είναι τα μητρώα αυτά δημόσια, είναι ένα ερώτημα, θα το αφήσω εδώ πέρα στην συνάδελφο. Για εμάς, για λόγους φορολογικούς, αρκεί να είναι διαθέσιμα στις φορολογικές αρχές. Αλλά αν είναι να μιλήσουμε για ένα ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον για την διαφθορά, θα μας απαντήσει η κυρία. Ε, να σου πω εγώ αν θα είναι λοιπόν, ε, αν θα πρέπει να είναι δημόσια. Η φορολογική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου τα τελευταία πέντε χρόνια έχει υποστεί μείωση του προπολογισμού της στο μισό. Ο αριθμός ε, των επιθεωρητών έχει μειωθεί στο μισό, οπότε έχουν αυξηθεί τα σχέδια φορολογικού επιθετικού σχεδιασμού. Οπότε όσο περισσότεροι τα βλέπουν αυτά, τόσο το καλύτερο. Ε, συχνά μάλιστα οι δημοσιογράφοι επισημαίνουν ε, πράγματα στην εφορία. Οπότε χρειάζεται πρόσβαση του κοινού γενικώ. Και οι τοπικές εφημερίδες πρέπει να ξέρουν τι συμβαίνει στον τόπο τους. Και οπωσδήποτε στο Ηνωμένο Βασίλειο εγώ έχω εργαστεί σε τρεις τέτοιες έρευνες και αυτό το οποίο βλέπω σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι μια πολιτική βούληση να ασχολούνται με υποθέσεις γνωστών ανθρώπων ε, για παραδειγματισμό. Παραδείγματος χάρη με την HSBC είχαμε τον πρόεδρο της ε, Santander ε, και η κληρονόμος της Νίνα Ρίτσι και τα λοιπά στην Ελβετία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε μία δίωξη ενό εργολάβου οικοδομών. Σε κάποιες χώρες δηλαδή δεν υπάρχει πολιτική βούληση να χρησιμοποιηθούν ε, οι εξουσίες που έχουν οι φορολογικές αρχές. Και αν όσα γίνονται γίνονται δημοσίως, τότε και το κοινό θα φροντίσει να υπάρξει εφαρμογή του νόμου. Όσον αφορά τα μητρώα, μια σημαντική παραδοχή είναι ότι χρησιμοποιούνται καταπιστεύματα για να κρυφτεί η ιδιοκτησία ε, και μάλλον έτσι θα υπονομευθεί το σύστημα των ε, μητρώων. Σας ευχαριστώ. Η Άννα Γκόμες από τους Σοσιαλδημοκράτες. Κύριε Πρόεδρε, <clears throat> ευχαριστώ. Πρώτα για τη Μάλτα. Στις περιπτώσεις SLAP, δηλαδή στρατηγικών αγωγών για να αποτραπεί η πληροφόρηση του κοινού. Είδαμε ε, δράσεις σλαπ κατά της Τάφνε Γαλήσια. Είδαμε ότι ελήφθη το OK του Πρωθυπουργού. Γιατί μίλησε και για τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό, η κυρία Γκάσταρη, προηγουμένω και τη στάση τη στην Βουλή των Κοινοτήτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι επιπτώσει του γεγονότο ότι υπάρχουν ε, σχέσεις μεταξύ ορισμένων εταιριών και της Cambridge Analytica που προσπάθησαν να βοηθήσουν να βοηθήσουν κάποια κόμματα να κερδίσουν εκλογές και όπως και σε κάποιες ε, υπερπόντιες βρετανικές κτήσεις. Είναι πολύ ανησυχητικό, το γεγονός ότι, ότι τα παιδιά και ο χείρος της ε, Γκαλίσια έχουν τώρα κληρονομήσει το εισαγωγικών όλες τις αγωγές. Έχουν φτάσει τώρα ε, τα πρόσωπα που έχουν λάβει χρυσές ε, βίζες τους 5.800. Μαζί όμως με τα, ε, με τα μέλη των οικογενειών φτάνουν τις 20.000 και οι περισσότεροι από αυτούς είναι οι Κινέζοι και δεν δίνει, δεν απολύτως καμία πληροφορία η κυβέρνηση. Υποτίθεται λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων, κάτι το οποίο ε, είναι απολύτως απογοητευτικό. Ερώτηση προς τον κύριο Πρόσ. Για τους πραγματικούς δικαιούχους είπε ότι για του η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η ε, διαφάνεια των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων δεν ε, αναμένεται διότι ε, δεν τα προβλέπει ο νόμος. Πότε θα γίνει όμως, πότε θα ισχύσουν τα πρότυπα του ΟΣΑ παγκοσμίω ώστε να ισχύσουν και εδώ. Και τι γίνεται όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι τραπεζικοί λογαριασμοί, είναι για παράδειγμα ε, ενσώματα αγαθά, τα οποία είναι ε, τοποθετημένα σε, ελεύθερες, σε ζώνες ελευθερών συναλλαγών. Για την κυρία Γκάρσαϊντ, μπορείτε να πείτε λίγα περισσότερα σχετικά με την αντίσταση που βλέπουμε από αυτά τα υπερπόντια εδάφη απέναντι στη Νέα Βρετανική νομοθεσία που επιτάσσει την δημοσιοποίηση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων, γιατί γίνεται μεγάλο λόμπι εναντίον. Και επίση για την Αμερικανική νομοθεσία που ίσω είναι χρήσιμη και για τι ευρωπαϊκέ δράσει. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Πρόσ, κύριε Γκασάιτ. Ευχαριστώ για τι θαυμάσιε ερωτήσει λέει ο κύριο Πρόσ, για την πρώτη σα για του πραγματικού δικαιούχου είναι μέγα θέμα. Είναι ζήτημα για την FADF, και ο ΩΣΑ θεωρεί, έχει περιλάβει μάλλον τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους στο πακέτο. Χρειάζεται λοιπόν, είναι, είναι φιλόδοξο το πρότυπο, αλλά η FATF αυτό που κάνει είναι ελέγχει τον βαθμό της εφαρμογής του προτύπου και στους G20 για παράδειγμα για να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε συνεπή εφαρμογή του προτύπου. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει. Έχουμε το πρότυπο. Είναι αναγκαίο να φροντίσουμε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. FATF και όσα δεν ζητούν να μάθουν πού βρίσκονται οι προφορίες, αλλά το πώς. Χρειάζεται παγκοσμίω να ισχύσει το πώς μπορεί να είναι καταχωρισμένο, αρκεί να είναι αποτελεσματικό. Και τέλος, είναι αναγκαίο να είναι δημόσιο κτήμα για την φορολογική κοινότητα, όχι. Για τους λογαριασμούς. Εάν δηλαδή αφαιρέσει κανεί τα χρήματα από το λογαριασμό και αγοράσει ας πούμε μια θαλαμιγό ή κοσμήματα ή κάτι άλλο. Είναι αληθέ ότι το σύστημα ανταλλαγών καλύπτει μόνο του χρηματοπιστωτικού λογαριασμού. Αν έχετε ένα πιστοποιητικό δηλαδή χρηματοπιστωτικού λογαριασμού. Δεν καλύπτονται λοιπόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Εάν ανακαλύψουμε λοιπόν ότι υπάρχει κάποια σημαντική διαρροή, πρέπει να το σκεφτούμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Τώρα, η εξισορρόπηση της υποχρέωσης υποβολής έκθεσης κλπ. Για να είμαστε ειλικρινεί, ακολουθήσαμε και το πρότυπο των ΗΠΑ. Βελτιώσαμε το σύστημα, βελτιώσαμε το Common Reporting Standard, καλύπτει ένα μεγάλο αριθμό περιουσιακών στοιχείων, όχι όμως όλα. Δεν έχουμε δηλαδή αυτόματο reporting για άλλα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό μπορεί να ζητηθεί αλλά ο αυτοματισμό αναφέρεται ειδικά στα στοιχεία των ε, χρηματοπιστωτικών λογαριασμών, τραπεζικών λογαριασμών δηλαδή. Η κυρία Γκάσάιντ. Πρώτον για τα υπερπόντια εδάφη. Και πού πάμε τώρα. Ο νόμος που ψηφίστηκε από το Βρετανικό Κοινοβούλιο και βεβαίως δεν έχει ικανοποιήσει πολύ την κυβέρνηση, διότι ήταν επανάσταση εντό αγωγικών κάποιων βουλευτών. Εάν τώρα η κυβέρνηση είναι πραγματικά σοβαρή για να, σε ό,τι αφορά την αλλαγή του καθεστώτος, ε, θα ανεγνώριζε ότι ε, χρειάζονται κάποιε μεταρρυθμίσει, α πούμε στις Βερμούδες, που βασίζονται πολύ σε αυτού του είδου τι ε, επιχειρήσει. Και χρειάζεται εκεί βέβαια και κάποιο πακέτο βοήθειας για να ενισχύσει τι οικονομίε των υπερπόντιων κτήσεων. Πρόκειται για εγκατεστημένα πρόσωπα εκεί που έχουν ε, μεγάλη εισοδηματική βάση. Τώρα, θα πρέπει να υπάρξουν δημόσια προσβάσιμα μητρώα. Βέβαια, δεν, η προσπάθεια αυτή δεν έχει πολύ μεγάλη δυνατότητα να επιτευχθεί, γιατί το κοινοβούλιο είναι κυρίαρχο. Και η κυβέρνηση θα πρέπει να υποστηρίξει την πολιτική αυτή. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα την υπερασπιστεί. Για τις στρατηγικές αγωγές για την αποτροπή της γνώσης του κοινού Υπάρχει νομοθεσία στι ΗΠΑ, δεν ξέρω ακριβώ πώ λειτουργεί. Προβλέπει όμω ποινέ. Και οι ποινέ αυτέ είναι αποτρεπτικέ. Είναι ούτω ή άλλω ε, και δαπανηρό να προσλάβει κάποιο ένα δικηγόρο ο οποίο θα πάει να κάνει μια αγωγή σλαπ. Δεν νομίζω όμως ότι μικρές εφημερίδες ή ε, ε, ε χαμηλούς δημοσιογράφοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους έτσι. Σε ένα λεπτό αρχίζει το επόμενο πάνελ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους, την κυρία Γκάσάιτ, την κυρία Ροσέλ, τον κύριο Προς. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Αλλάζει τώρα το σκηνικό και συνεχίζουμε στις 10.40 ακριβώς με το επόμενο πάνελ. Ο Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, ας αρχίσουμε τώρα ε, το δεύτερο πάνελ. Well, so, dear colleagues, we will resume our, our... Αυτή την δημοσία ακρόαση με το δεύτερο σε σχέση με αυτές τις ε, επιθετικές, επιλήψιμες φορολογικές πρακτικές όσον αφορά το τι γίνεται στην ε, Ευρώπη. Όπως σας είπα στην ε, αρχή της ακροάσεως, μίλησαμε για τις πολυεθνικές που είχαμε προσκαλέσει στην ακροασή μας. Και τώρα Καλώς όρισαν η κυρία Irene Yates που είναι αντιπρόεδρος της ε, υπηρεσίας της McDonald's για τον ε, εταιρικό φόρο και την κυρία Πατρίσα Τζόνσον που έχει την αντίστοιχη θέση στην Nike. Η καθεμία έχει στη διαθεσή της 10 λεπτά για την εισήγηση. Οπότε παρακαλούμε κυρία Γέιτς. να μας κάνετε την εισήγησή σας. Σας ευχαριστώ και καλημέρα. Ευχαριστώ που σήμερα με καλέσατε για να βοηθήσει η συζήτησή μας να σας δώσω και επιστήμες πληροφορίες για την McDonald's. Στην Ευρώπη έχουμε δραστηριότητα σε 39 χώρες και σε όλα τα κρατημέλη, πάνω από 8.000 εστιατόρια. 15 εκατομμύρια είναι πελάτες μας στην Ευρώπη κάθε μέρα και απασχαλούμε 425.000 και πάνω υπαλλήλους. 90% ε, ε, από τα υλικά μας προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Γεωργία και έτσι βοηθούμε την Ευρωπαϊκή Οικονομία. Έχουμε κάποια πρωτοτυπία σχέση με άλλες μεγάλες εταιρείες γιατί η εταιρεία μας στηρίζεται σε ένα franchise. Πάνω από 85% των εστιατορίων μας είναι με το σύστημα franchise από ανεξάρτητους επιχειρηματίες και γυναίκες. Ε, αυτό διότι ωφελούνται πάλι από αυτό το σύστημα, μπορούν να αναπτύξουν την επιχείρησή τους και μακρόπνο και έχουν επομένως τη σχετική άδεια για την λειτουργία των McDonald's που έχουν. Και είναι καινοτόμο το σύστημα, διατροφική ασφάλεια, στο design, όσον αφορά τη μεταχείριση των ε, ε, καταναλωτών. Είναι ανεξάρτητοι επομένω επιχειρηματίε και καταβάλουν κάποιο δικαίωμα για το δικαίωμα το οποίο έχουν ούτως ώστε να χρησιμοποιούν το σύστημα μας και έτσι μπορούμε να επενδύσουμε, μπορούμε να αναπτυχθούμε ε, προς την καινοτομία και το ποσόν αυτού του δικαιώματος υπολογίζονται προσεκτικά σύμφωνα με τα εργαλεία του ΟΣΑ. Είναι δίκαιο το το πρέπει να πληρώνουν σύμφωνα με τις αρχές που διέμουν την αγορά επίσης. Τώρα, όσον αφορά τα φορολογικά, πληρώνουμε σημαντικά ποσά σε εταιρικό φορά στην Ευρώπη. Και επίσης ε, πληρώνουμε και τις κοινωνικές εισφορές κλπ. Από το 2013 με το μέχρι τις 2017 δώσαμε πάνω από 3 δις δολάρια σε εταιρικού φόρους. Και ο μέσος ήταν 29%. Και πληρώνουμε και φόρου κοινωνική πολιτικής και άλλους. Και πάρα πολλέ ε, εταιρείε έχουν έδρα εκεί που δρούν και υπάγονται στο δίκαιο αυτών των χωρών και πληρώνουν το φόρο σε αυτές τις χώρες. Οπότε και οι επιχειρηματίε που αναλαμβάνουν τα McDonald's επίση πληρώνουν εταιρικό φόρο και Επομένω, είναι σημαντικό ο φως που στην Ευρώπη. Το 2015 είπαμε ότι θα αναδιοργανωθούμε και στη συνέχεια είπαμε ότι θα έχουμε ένα καινούριο επιχειρηματικό μοντέλο. Η αλλαγή αυτή οδηγήσε σε μια ενιαία δομή στο Ερμηνο Βασίλειο και από εκεί υπήρχε αρμοδιότητα για να δίνονται τα ε, δικαιώματα πραγματικής διοκτησίας παντού εκτός από τις ΗΠΑ και έτσι είχαμε καλύτερη δομή λήψης αποφάσεων, καλύτερη υποστήριξη του franchise. Και οπότε κλείσαμε το κέντρο το επιχειρηματικό μας στην Γενέβη. Ε, βέβαια στο Κρισιέ παραμένουν τα γραφεία μας και συνεχίζουμε να έχουμε το γραφείο μας στο Λουξεμβούργο για τα εκεί εστιατόρια. Έχουμε πολλούς ε, υπαλλήλους στο Λονδίνο. Γι' αυτό διαλέξαμε αυτό ως κέντρο. Έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό, ε, λόγω της γλώσσας, λόγω των διασυνδέσεων με άλλες αγορές και αποφασίσαμε να αναδιοργανωθούμε και να ευθυγραμμιστούμε με τα δεδομένα του ΟΣΑ και το BEPS ε και τα Paradise Papers. Τι χρειάζεται. Χρειάζεται να είναι ξεκάθαρη νομοθεσία. Αυτό θέλει κάθε επιχείρηση, κάθε εταιρεία. Και να είναι ξεκάθαρο και το φορολογικό καθεστώς. Ξεκάθαρε κατευθυντήριε. Έτσι η φορολόγηση είναι πιο συνεπής. Για τον BEPS θέλουμε να γίνεται μια σφαιρική και όχι αναχώρα εφαρμογή του BEPS. Υπάρχει ασφαλεία δικαίου, για τα φορολογικά. Αυτό θέλει η εταιρεία. Ασφάλεια δικαίου, συνέπεια και κάθε κατάσταση για κάθε νέο νόμο. Έτσι μπορεί η εταιρεία να συνεχίσει την αναπτύξή τη, να δημιουργεί θέσει απασχόληση και να πληρώνει εκεί που πρέπει, εκεί που δρά ε, στην Ευρώπη και παντού. Σε ευχαριστώ και περιμένω πώς και πώς τη ζήτησή μας. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γέιτς. Τώρα θα ακούσουμε την κυρία Τζόνσον. Καλημέρα σας, λέγομαι Πατρίσια Τζόνσον. Είμαι η Διευθύντρια Φορολογικής Πολιτικής της ΝΑΕΚΙ. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την ευκαιρία αυτή που μας δίνετε για να συζητήσουμε μαζί σας το πώς οργανώνουμε την επιχείρησή μας και να συνεισφέρουμε σε έναν επικοδομητικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα θα ήθελα να τονίσω δύο πτυχές της επιχειρήσή μας. Πρώτα απ' όλα συμβάλλουμε σημαντικά στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό γίνεται μέσω των επενδύσεών μας, των θέσεων εργασίας που δημιουργούμε, της καινοτομία και βεβαίως μέσω του πάθους για τον αθλητισμό που προωθούμε. Δεύτερον, όσον αφορά τη φορολογική πολιτική, παρακολουθούμε τις εξελίξεις για δύο βασικούς στόχους, για να προσαρμοστούμε, για να ακολουθούμε τους παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς φορολογικούς κανόνες, κυρίως τις αλλαγές κατευθύνες γραμμές του ΩΣΑ και να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους της κάθε χώρας στην οποία λειτουργούμε. Ως μια εταιρεία με παγκόσμιες λειτουργίες θέλουμε μια φορολογική πολιτική η οποία θα ευνοεί το επιχειρηματικό κλίμα, θα είναι απλή και συνεπής στην παγκόσμια εφαρμογή της. Έτσι θα μπορούμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε με εμπιστοσύνη και να εμπνέουμε τη σημερινή και την αυριανή γενιά αθλητών. Η Nike είναι έχει εμπλακεί σε μακροχρόνιες επενδύσεις στην Ευρώπη. Από του 74.000 υπαλλήλου μας έχουμε πάνω από 14.000 υπαλλήλου σε 20 χώρες στην Ευρώπη. Είμαστε παρόντες στην Ευρώπη από το 1972 και με κλίμακας επιχειρήσεις από το 1987. Από το 1998 τα κεντρικά μας στην Ευρώπη βρίσκονται στο Χίλβερσουμ τη Ολλανδία, όπου απασχολούμε 2.500 ανθρώπου. Επιλέξαμε την Ολλανδία για πολλού λόγου. κυρίω την γεωγραφική της, την κεντρική γεωγραφική της θέση, το γεγονός ότι έχει πολύ καλούς εργαζομένους και ένα δυναμικό αλλά σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Επίσης έχουμε ένα παγκόσμιο κέντρο διανομής στο Βέλγιο που απασχολούμε 3.500 άτομα. Οι επενδύσεις μας στους ανθρώπους, στο marketing, σε ακίνητα, σε ε, σε οργάνωση επιμελητίας και η συνεργασία μας με πάνω από 7.500 μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι απόδειξη του πόσο προσιλωμένοι είμαστε στην Ευρώπη. Η έδρα μας είναι στο Beaverton, Oregon και δουλεύουμε μέσω δύο διάβλων, της χοντρικής πώληση και της άμεσης πώληση λιανικής στους καταναλωτές. Έχουμε λοιπόν 309 ιδιόκτητα καταστήματα στην Ευρώπη και συνεργασία με 5.500 καταστήματα χοντρικής και όλο και περισσότερο μέσω της ψηφιακής οδού. Η καινοτομία μας και η ανάπτυξη προϊόντων γίνεται κυρίως στη ΣΥΠΑ. Η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει εμπορικά σήματα και ε, πατέντες, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για το για την ε, εταιρεία μας, την επιτυχία μας και την ανταγωνιστική μας ε, θέση. Η επιχειρηματική μας δομή αντικατοπτρίζει τις πραγματικότητες και την ζήτηση της παγκόσμιας οικονομίας και βρίσκεται σε πάρα πολλές χώρες, έχει πολλές γραμμές παραγωγής ε, και διάβλους διανομής. Η φορολογική μας δομή επίσης αντικατοπτρίζει την επιχειρηματική μας δομή. Στόχο έχει να διευκολύνει την παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών με τον πιο αποτελεσματικό και φτηνό τρόπο στους πελάτες μας η φορολογική μας δομή συμμορφώνεται με την διεθνή νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΩΣΑ και το ευρωπαϊκό δίκαιο και τους νόμους των χωρών όπου λειτουργούμε. Θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα γεγονότα εδώ. Το 2017 η φορολογική μας δαπάνη στην Ευρώπη που περιλαμβάνει και φόρους ε, στην μισθοδοσία και στην ιδιοκτησία και φόρο επιχειρήσεων ήταν πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο του 2018 με τις αλλαγές στην Αμερικανική νομοθεσία είχαμε φορολογική δαπάνη σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα συσσωρευμένα κέρδη στο εξωτερικό. Οπότε όλα τα παγκόσμια κέρδη της Nike φορολογούνται. Αναγνωρίζουμε πως οι διεθνείς φορολογικοί κανόνες αλλάζουν σύνεχώς και η εταιρεία πάντα προσαρμοζόταν και θα συνεχίσει να προσαρμόζεται στις αλλαγές για να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους κάθε χώρα στην οποία λειτουργούμε. Εν ολίγης, ελπίζω τα σχόλια αυτά να συνεισφέρουν σε έναν επικοδομητικό διάλογο με την Ειδική Επιτροπή σας και την παγκόσμια οικονομία. Και είμαι στην διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ξεκινάει τώρα η συζήτηση και πάλι θα γίνουν ερωτήσεις ε, σε 5 λεπτά διαστήματα, ένα λεπτό η ερώτηση και 4 λεπτά η απάντηση. το ΕΛΚΟ, κύριος Νίντερμαϊρ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτιμώ την παρουσία σας, κυρίες μου, γιατί ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να έρθετε σε μια κρόάση και να μας μιλήσετε. Κάποιες εταιρείε αποφάσισαν να μην ε, έρθουν και θέλω να πω ότι εκτιμώ ιδιαιτέρως τις ερωτήσεις σας και δεν θα ασχοληθώ συγκεκριμένα με τα φορολογικά σας. Θα ήθελα να μιλήσω ευρύτερα. Έχω την εντύπωση ότι τις τελευταίες δεκαετίες πολλές εταιρείες αφιέρωσαν πάρα πολλούς πόρους στην βελτιστοποίηση ε, των φορολογικών συστημάτων αντί για την βελτιστοποίηση του προϊόντος. Και κάποιες είναι πολύ επιτυχείς, οφείλω να πω. Και η συνέπεια είναι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι και οικονομολόγοι και πολιτικοί δεν θεωρούν ότι είναι βιώσιμη η φορολογική κατάσταση που έχει αναπτυχθεί γιατί δεν είναι δίκαια. Μπορούμε να πούμε ότι ο φόρος θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το πού βγάζουν τα κέρδη οι εταιρείε ε, και πλέον υπάρχει μια πλήρης αποσύνδεση μεταξύ της δημιουργίας των κερδών και το πού πληρώνουν οι εταιρείε φόρο. Δεν θέλω να υποτιμήσω οπωσδήποτε τα ζητήματα φορολογίας πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιόχρησης ε, και τα λοιπά. Πράγματι υπάρχει εδώ ένα περιθώριο, αλλά ε, όλοι θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξουν οι υφιστάμενες ε, πρακτικές. Η κοινωνία προφανώς απαιτεί περισσότερη διαφάνεια και σε τελική ανάλυση να δούμε δηλαδή και το αποτέλεσμα. Όταν ε, έχετε κέρδη πρέπει να πληρώνετε και κάποιους ε, φόρους. Βεβαίως ε, τα μέτρα θα είναι νομοθετικά αλλά και μη νομοθετικά, πειθώ. και βεβαίω ζητήματα κοινωνικής ευθύνη των εταιριών. Οπότε η ερώτησή μου είναι εξή: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει κάποια ανάγκη να αλλάξουν οι επιχειρήσει σα, αν έχετε δει κάτι τέτοιο τα τελευταία πέντε χρόνια και... Οι Και βεβαίω ε, αν μπορείτε να μα πείτε, αν διαφέρουν οι πρακτικέ αυτέ από τη μία εταιρεία στην άλλη. Σα ευχαριστώ. Ποια θα ήθελε να απαντήσει. Ναι, παρακαλώ εσεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, ερώτησή σας. Όπως είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, τα McDonald's έχουν πληρώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε φόρους σε ολόκληρη την Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια. Ε, εταιρικούς φόρους. Εμείς ως εταιρεία, όπως είπε και η Nike, έχουμε μια εταιρική δομή και φορολογική δομή που ακολουθεί το επιχειρηματικό μοντέλο, δεν ε, το καθοδηγεί. Οπότε οι αλλαγέ που κάναμε και οι πιο πρόσφατες μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο στην εταιρεία μας εκεί ήταν ως αποτέλεσμα του νέου διευθύνοντος συμβούλου που άλλαξε την δομή από γεωγραφική σε κλαδική, σε τμήματική. Οπότε αυτά τα ακολουθεί η φορολογική πολιτική μας, δεν τα καθοδηγεί. Πληρώνουμε τους εταιρικούς φόρους σε κάθε χώρα που έχουμε εστιατόρια, τα εστιατόρια λειτουργούν τοπικά και εκεί πληρώνουμε το φόρο. Η κυρία Τζόνσον. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ευχαριστώ και την Αγία που απάντησε πρώτη. Να πω ότι και εγώ από την εμπειρία μου με την Nike δεν έχουμε μεταφέρει τις επιχειρήσεις μας για να κατασκευάσουμε τα φορολογικά αποτελέσματα. Τα φορολογικά ε, παρακολουθούν και διευκολύνουν την διεξαγωγή των ε, επιχειρήσεών μας. Μάλιστα. Ο συνεισηγητής για τους σοσιαλδημοκράτες, ο κ. Σκοφότη. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας ε, για να απαντήσετε ερωτήσεις. Εγώ θα περιοριστώ στην ε, κυρία Γέιτς. Από το 2015 έως το 2018 McDonald's ε, έχει αλλάξει δραματικά την εταιρική δομή της. Σύμφωνα με την έκθεση Unhappy Meal, ε, που ίσως ξέρετε, οι δραστηριότητες ε, της McDonald's το 2015 ελέγχονταν από 6 εταιρίες με έδρα της ΙΠΑ και το Λουξεμβούργο. Σήμερα όμως χρειάζεστε 11 εταιρίες με έδρα ΙΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κόνγκ και Ολλανδία και μιλήσατε για την ανάγκη σαφήνειας. Οπότε η πρώτη μου ερώτηση είναι ποιος είναι ο συγκεκριμένος ε, λόγος ε, ή λόγοι για τις ε, αλλαγές αυτές και την περιπλοκότητα στις δομές σας. Και δεύτερον, όσον αφορά την πρόσβαση σε προσοντούχους εργαζομένους. Η απόφασή σας να φύγετε από το Λουξεμβούργο σχετίζεται με την έρευνα της ε, Κομισιόν για τα φορολογικά του Λουξεμβούργου ή στην ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου για, τον χαμηλότερο, για τη χαμηλότερη φορολογία επιχειρήσεων. Πέρα δηλαδή από το προσοντούχο προσωπικό. Σας ευχαριστώ, έχετε τον λόγο. Θα ξεκινήσω από την ε, τελευταία ερώτηση. Η απόφαση της εταιρείας να μετακινηθεί από το Λουξεμβούργο στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε ακριβώς το ότι η δομή μας άλλαξε και μεταφέρθηκε σε τμήματα. Δηλαδή οργανώσαμε ε, πέντε χώρες ε, που έχουν ηγετικό ρόλο και ουσιαστικά είναι το 40% των εσόδων μας κοιτώντας ε, και αναζητώντας τρόπους να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στην λήψη αποφάσεων ε, και τον διαμοιρασμό πληροφοριών, σκεφτήκαμε πού ήταν το καλύτερο μέρος για να γίνει αυτό και το Ηνωμένο Βασίλειο προέκυψε καθώς ήταν κοντά στις άλλες αγορές, είχε γλωσσικές ομοιότητες με τη μητρική εταιρεία στη ΣΥΠΑ και όπως είπατε είχε και πρόσβαση σε προσοντούχους ανθρώπους. Υπήρχε λοιπόν μια βάση εκεί ήδη. Η ανάλυση της απόφασης ε, είχε προηγηθεί του Brexit ε, και τις ανακοινώσεις του ΟΣΑ του Ιουνίου 17 και των Paradise Papers και δεν ε, είχε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή κρατικών ενισχύσεων και εκτιμάτε εσείς ε, την συμμετοχή μας ε, και ε, θα μου επιτρέψετε και εμένα να μην σχολιάσω σε έρευνες οι οποίες ακόμα εκκρεμούν. Οπότε δεν σχετιζόταν. Θέλετε να επανέλθετε. Όχι, όχι, ναι, δεν το ξέχασα. Όσον αφορά τις αλλαγές στη δομή μας αυτό το οποίο έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το αποτέλεσμα μιας μετάβασης σε κάποιες ε, περιπτώσεις για νομικούς λόγους. Μετακινήσαμε μια ε, εταιρεία αντί να γίνει μόνο μια μετακίνηση στη ενεργητικών. Λοιπόν, αυτό οδηγεί και σε διοικητική απλότητα, παραδείγματο χάρη λιγότερα συμβόλαια δικαιόχρηση. Κάποιου από τους ε, κανόνε μα οδήγησαν να επιλέξουμε τη μία χώρα έναντι της άλλης. Αλλά για να γίνει αντιληπτό το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν ζητήσαμε ούτε λάβαμε ειδική μεταχείριση φορολογική του Ηνωμένου Βασιλείου. Πληρώνουμε πλήρη φόρο στο καθαρό κέρδος, ναι. Ίσως δεν ακούσατε καλά την ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση ήταν ο συγκεκριμένος λόγος ε, για τις πολύπλοκες αλλαγές στην εταιρική δομή σας στην Ευρώπη, όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά το ότι χρειάζεστε 11 εταιρείε με έδρα ΙΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Σιγκαπούρη και αλλού. Δηλαδή περάσατε σε ένα πολύπλοκο σύστημα εταιρική ε, δομή και δεν αντιλαμβάνομαι τον λόγο. Είναι για φορολογικούς λόγους ή για κάποιον άλλο λόγο. Όχι, δεν είναι για φορολογικούς λόγους. Ε, δεν έχουμε έδρα καθόλου στην ε, Ολλανδία. Έχουμε 75 εστιατόρια, ε, δικαιούχους δηλαδή, δικαιόχρησης. Ε, τώρα δεν είμαι σίγουρη ότι η έκθεση αυτή την οποία αναφέρατε είναι 100% ακριβής. θα ήθελα εγώ να εστιάσω στο εξή. Αν σκεφτείτε το που ήμασταν πριν, έγινε μια μετάβαση, δηλαδή είχαμε περιφερειακή έδρα στην Σιγκαπούρη. Αυτή μετακινήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, αν μου επιτρέπετε, κυρία Γκέιτς, είπατε ότι δεν είναι σωστές όλες οι πληροφορίες της έκθεσης. Μπορείτε να μας δώσετε μια γραπτή απάντηση για το τι δεν είναι ακριβές στην έκθεση αυτή, για να δούμε τι είναι σωστό και τι λάθος. Ε, όχι, δεν βλέπω κάποιο λόγο για αυτό. Ε, αυτό το οποίο εμείς κάνουμε ως μια υπεύθυνη εταιρεία είναι ότι έρχομαι εγώ να σας πω τι συμβαίνει ακριβώς. Ναι, ναι, επειδή μιλάτε για σαφήνεια, θα θέλαμε και η Επιτροπή να λάβει ε, το τι θεωρείται ανακριβές στην έκθεση αυτήν. είναι κάποια στοιχεία ανακριβή, επειδή είπατε ίδια ότι είναι ανακριβή. Το, εγώ το απάντησα, δεν, δεν βλέπω το λόγο να σας δώσω τις πληροφορίες. Ευχαριστώ να απαντήσω στις ερωτήσεις που συζητάμε. Κύριος Φανκάντελαρε, καλημέρα σας ε, κυρία Γέιτς. Ε, Είχα χθες το βράδυ, έφαγα σε ένα εστιατόριό σας και άρα δεν ε, σκώ μόνο για να ασκήσω κριτική αλλά στην γραπτή σας απάντηση μιλάτε για την αναδιοργάνωση από το 2015 και βλέπουμε ότι αυτή η αναδιοργάνωση ε, έλαβε χώρα πρώτα απ' όλα μετά το ξεκίνημα έρευνας για τα Lux Leaks από την ε, Κομισιόν και την υπογραφή από τη ΣΥΠΑ της ε, Σύμβασης ε, για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας και βεβαίως και ακριβώς συνέπεσε με το Brexit το 2016. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με σύμπτωση. Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα ζήτημα αντίληψη όταν αρχίζετε να αλλάζετε την επιχειρηματική σα δομή ακριβώ τη στιγμή που ξεκινάει μια έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερη ερώτηση. Ε, δεδομένη τη ε, αναθεώρηση ε, τη ε, Σύμβαση Αποφυγή Διπλή Φορολογία ή Λουξεμβούργου έπαιξε και αυτό έναν ρόλο και κάτι άλλο για την επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου. Είπατε στην ε, εισαγωγή σας ότι ελήφθη η απόφαση ε, για λόγους ε, προσοντούχου, προσωπικού και πως ήταν και αυτός ένας λόγος για να πάτε στο Λουξεμβούργο και εκεί πέρα ήταν το ίδιο το ζήτημα γλώσσας και προσωπικού. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γέιτς. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Στις εναρκτήριες παρατηρήσεις μου σας εξήγησα ότι η απόφαση της εταιρεία να κάνει αναδιάρθρωση έγινε γιατί αλλάξαμε το επιχειρησιακό μας μοντέλο, γιατί είχε αλλάξει το Μάρτιο του 15 ο Διεθνών Σύμβουλος, οπότε και ε, έτσι εξηγείται αυτό που είπατε αν είναι ε, σύμπτωση. Είναι. Δεν έχει σχέση με τις ε, ε τότε έρευνες που άρχισαν. Αυτά όσο εξήγησε. Και τώρα όσον αφορά το γιατί επελέγει το Ηνωμένο Βασίλειο ως έδρα, ως κέντρο για την παροχή των αδειών franchise κλπ. Είπαμε ότι αυτό έχει να κάνει με, τη, με τα αγγλικά ως γλώσσα εργασίας κλπ. Σχέση με άλλες αγορές. Οπότε η απόφαση για το Λουξεμβούργο ελήφθη το 2009. Ε, αυτό έγινε επί τη βάση άλλου επιχειρηματικού μοντέλου και σας παραλαμβάνω ότι αυτό το οποίο κάνουμε τώρα είναι ότι εφαρμόζουμε ένα τέτοιο παγκόσμιο μοντέλο επιχειρηματικό με προσανατολισμό προς την κοινοτομία σε αλλαγές που να καλύπτει αυτό το μοντέλο το εστιατοριά μας όπου να πτήσουμε επιχειρηματική δραστηριότητα. επιτρέπετε άλλη μια ερώτηση είναι σημαντική η καινοτομία για σας. Θεωρείτε ότι μπορεί να αποτελέσει και η διαφάνεια μέρος της καινοτομίας. Δεν, δεν άκουσα το τέλος ότι σας είπα κατά πόσον και η διαφάνεια είναι κομμάτι της προσπάθειάς σας για καινοτομία. Α, αυτό, αυτό, μετά, μετά το είπατε. Η κυρία συνεχίζει. Ναι, έχουν τολισμό τέτοιο για την ε, διαφάνεια και την καινοτομία και εστιαζόμαστε στην λειτουργία των εστιατορίων στο μενού, στο design, την τεχνολογία, στο να φουγκραζόμαστε τους πελάτες. Διαφάνεια τώρα από πλευρά εταιρικού φόρου. Αυτό σημαίνει ότι συμμορφωνόμαστε με το φορολογικό δίκαιο, ότι καταβάλουμε το φόρο εκεί όπου αναπτύσσουμε δραστηριότητα, ε, υποβάλλουμε τις αναφορές εκθέσεις που προβλέπονται και πληρώνουμε ένα σωρό φόρο εκεί όπου ε, αναπτύσσουμε δραστηριότητα. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος Σίμων. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή μου θα διατυπωθεί στα γερμανικά, παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά. Θα έλθω ξανά σε αυτό που είπε ο κύριο Κόφουτ. Και σα παρακαλώ κυρία Γίτ. αν θέλετε να κοιτάξετε προς το μέρος μου. Είμαι εδώ πίσω σας δεξιά. Α, εδώ. Έχω εδώ μια έκθεση που ονομάστηκε το μη ικανοποιημένο γεύμα, το unhappy meal και δείχνει την εταιρική δομή των McDonald's πριν από την εγκατάστασή του στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά. Πριν βλέπει κανείς μια ξεκάθαρη γραμμή και μετά βλέπει κανείς, μετά δηλαδή από αυτή την κίνηση, μια, ένα πλήθος διασυνδεωμένων επιχειρήσεων. Μπορείτε να εξηγήσετε με απλά λόγια σε έναν απλό άνθρωπο τον λόγο που να μην είναι αδιαφάνεια, για ποιο λόγο περνάτε από μια ξεκάθαρη δομή με μια αναδιάρθρωση σε ένα σύστημα που νομίζω ότι καμιά φορολογική αρχή πλέον δεν θα μπορέσει να ξεδιαλύνει. Ο Πρόεδρος, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους κάνα την αδιάθρωση, εάν δεν πρόκειται για φορολογικού λόγους. Η κυρία ε, Γέιτς. Όπως είπα, υπάρχει ένας αριθμό λόγων νομικών για τους οποίους έχουμε μετακινήσει στοιχεία ενεργητικού και εταιρείε με ε, τελική, τελικό σκοπό την εγκατάστασή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτι που είναι σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό, είναι ότι πληρώνουμε τους φόρους που μας αναλογούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχουμε ούτε ζητήσει ούτε λάβει ή κίνητρα ή ειδικέ φορολογικές αποφάσεις. Έχουμε μια σημαντική επιχειρησιακή βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουμε και τα δικαιώματα για πάνω από την μισή διανοητική ιδιοκτησία εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Εσείς κύριε Σίμων τώρα, ας το αφήσουμε αυτό, γιατί δεν υπάρχει και τόσος χρόνος, να δούμε κάτι άλλο. Έχετε δώσει γραπτές απαντήσεις, τις οποίες αναφέρεστε στα κριτήρια του ΟΟΣΑ σχετικά με τα δικαιώματα που πληρώνονται για τις άδειές σας και την αρχή arm's length, δηλαδή την ανεξαρτησία αγοραστού πολιτού. Μπορείτε να μου εξηγήσετε αυτή την αρχή arm's length, πώς την εφαρμόζετε. Η μάρκα McDonald's είναι μοναδική στο, στο ε, παγκοσμίω. Ποια κριτήρια χρησιμοποιείτε για τους εσωτερικούς ε, λογιστικούς συμψηφισμούς που κάνετε μέσα στην επιχείρησή σας για τα διάφορα των διαφόρων δικαιωμάτων και για την δικαιόχρηση που εκχωρείται. Απάντηση. Η McDonald's συμμορφώνεται με την νομοθεσία διαμόρφωσης των τιμών και επίσης και για την πληρωμή, για την καταβολή δικαιωμάτων που ωφελούν τους ε, δικαιούχους δικαιόχρησης και αυτά αφορούν την μάρκα McDonald's τις ε, δομές και Υπάρχουν, υπάρχουν διαφορετικές δυναμικές σε διάφορες αγορές, αλλά γενικώ χρησιμοποιούμε μεθόδους διαμόρφωσης των τιμών ερεχόμενες όπου αυτές είναι διαθέσιμες, και ως οργάνωση franchise η McDonald's είναι διαφορετική από μεγάλες, άλλες μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Έχουμε πάνω από 85% των επιχειρήσεών μας των δραστηριοποιήσεών μας δηλαδή στην, στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, με αδειοδοτήσεις εστιατορίων. Κάνουμε και μια προσπάθεια franchising παγκοσμίω για να φτάσουμε στο 95% κάτι το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 350 εστιατόρια σήμερα που διαχειρίζεται η McDonald's γιατί είμαστε παγκόσμια εταιρεία στο 90% δηλαδή των χώρων. Διασφαλίζουμε transfer pricing κατάλληλο και βέβαια και κατάλληλα δικαιώματα. Max Anderson, Queens. Thank you. And thank you to αντεσο Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα πρώτα ήλθατε εσεί, κύριε Γέιτ, εκπρόσωπε του McDonald's, ενώ άλλοι όπως Apple δεν ήρθε καθόλου. Ω γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να ε, νομοθετήσει σχετικά με την υποβολή εκθέσεων αναχώρα για να ενισχύσει τον αγώνα κατά τη φορά αποφυγής. Αυτό θα γίνει όταν κάποιε χώρε μέλη και το Συμβούλιο και δυστυχώς και η Σουηδία όπου είναι πολύ δύσκολοι σοσιαλδημοκράτε, σταματήσουν να μπλοκάρουν. Θα γίνει όμως. Έχετε κάποια προβλήματα με την φήμη σα, λόγω φορολογικών θεμάτων και διαρωτώ με εάν θα ήσασταν διατεθειμένοι για να ενισχύσετε την φήμη σα, να αρχίσετε ήδη με την εφαρμογή των δημοσίων εκθέσεων αναχώρα ώστε να γνωρίζουν, να γνωρίζουν όλοι πού ε, αποκομίζεται κέρδος και πού πληρώνεται φόρους, εάν πληρώνετε φόρους. Σε ό,τι αφορά τη McDonald's, πολύ καλά κάνετε και πληρώνετε τους φόρους που δεν μπορείτε να αποφύγετε. Η δική μου ανησυχία είναι ωστόσο ότι έχετε μια πολύ περίπλοκη εταιρική δομή που σας διευκολύνει να μην πληρώσετε άλλους φόρους. Θα σας ρωτήσω συγκεκριμένα για την κίνηση του franchising από το Λουξεμβούργο στο, στην πολιτεία Delaware των ΗΠΑ. Η Delaware είναι δικαιοδοσία με πολύ περιορισμένες απαιτήσει ε, δημοσιοποίησης. Αυτό κατά κάποιο τρόπο επηρέασε την απόφασή σας για την Nike. Σύμφωνα με τα Paradise Papers έχετε μεταφέρει πολλά χρήματα από και προς την, τις Βερμούδες στην θηγατρική ε, της, ε, των Βερμούδων που έχουν μηδενικό συντελεστή, μηδενικό φορολογικό συντελεστή. Μπορείτε να μας πείτε πόσους ε, εργαζομένους έχετε επί του παρόντος στις Βερμούδες. κυρία Γέιτς, η πολιτεία Ντελαγουέα έχει ένα εξαιρετικό σύστημα φορολογία στις ΗΠΑ και ιδίω για, για την εταιρική φορολόγηση. Έχει και ιδιαίτερη ευκαμψία σε ό,τι αφορά την ε, η νομοθεσία τη, δηλαδή για την ίδρυση επιχειρήσεων. Πάνω 50% των επιχειρήσεων στι ΗΠΑ έχουν γίνει, έχουν ιδρυθεί στην πολιτεία Delaware και αυτό δεν έγινε για να αποφύγουν την φορολογησή τους οπουδήποτε. Εγώ να απαντήσω για τις Βερμούδες. Ε, υπό την Αμερικανική φορολογική νομοθεσία έχουμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε φόρους και δικαιώματα που εισπράττονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι ότου επαναπατριστούν στις Ηνωμένε Πολιτείες. Έχουμε δύο δισεκατομμύρια φορολογική επιβάρυνση για εξωτερικά έσοδα. Έχουν πληρωθεί οι φόροι δηλαδή για όλα τα έσοδα που έχουμε συλλέξει στις Βερμούδες και που επαναπατρίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορώ να απαντήσω και στην ερώτησή σας για την έκθεση αναχώρα. Απαντήσαμε ήδη γραπτός ότι οι εκθέσεις αυτές ε, κοινοποιούνται σε αλλοδαπές φορολογικές αρχές, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο ΩΣΑ και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά και η Αμερικανική Νομοθεσία. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε τις σχετικές εκθέσεις. Ο ΩΣΑ κατά επανάληψη έχει επιβεβαιώσει ότι οι εκθέσεις αυτές χρησιμοποιούνται μόνο από φορολογικές αρχές και μόνο για τον, την αξιολόγηση του κινδύνου. Μπορείτε να χθέσετε και μια ε, ερώτηση, follow-up κύριε Άντερσον. Πολύ σύντομο για την ε, εκπρόσωπο της εταιρείας McDonald's δεν αρνίζεται το γεγονός ότι η πολιτεία Delaware έχει πάρα πολύ περιορισμένες ε, απαιτήσει δημοσιοποίησης και μου λέτε απλώς ότι και όλοι οι άλλοι το κάνουν το ίδιο. Μήπως μπορείτε να απαντήσετε και εσείς στην ερώτηση για την ε, κοινοποίηση των εκθέσεων αναχώρα. Είχε δύο σκέλη η απάντησή μου για την πολιτεία Delaware. Είπα ότι πρώτον δεν είναι ασύνηθες κάτι τέτοιο για μια αμερικανική επιχείρηση να έχει την έδρα της Delaware. Κυρίως όμως λόγω του δικαστικού της συστήματος η Delaware έχει κρατική φορολογία, οι φόροι υποπληρώνονται στη Delaware. Σε ό,τι αφορά την έκθεση αναχώρα, θα συμφωνήσω με την κυρία Τζόνσον ότι ασφαλώς και συμμορφούμεθα με τον νόμο, υπάρχουν ισχυροί λόγοι και διεξάγονται συζητήσεις σχετικά με το πώς θα πρέπει να κοινοποιούνται οι εκθέσεις αναχώρα και επί του παρόντος αυτό που απαιτείται είναι να κοινοποιούνται στις φορολογικές αρχές και αυτό πράττει και θα συνεχίσει να πράττει η McDonald's. Πρόεδρος, υπενθυμίζω ότι η προηγούμενη εξεταστική επιτροπή Πάναμα είχε επισκεφθεί και την Τελαγουέα και είχαμε δει την κατάσταση σε μια αποστολή επιτόπου. Τώρα η κυρία Παλώμα Λόπες από την Ενωτική Αριστερά. Θα επιβάλλω την ερώτησή μου στα Ισπανικά πρόεδρα. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν επιθετικές φορολογικές θετικές στα κράτη ούτως ώστε να υπάρχει ελκυστικότητα για τι Τώρα έχουμε καλέσει τρει επιχειρήσεις που είναι κατά κάποιο τρόπο ε, άριστε, πρωταθλήτριε σε αυτό το τομέα. Ναι, δεν είναι βέβαια παράνομο, αλλά δεν ξέρω αν είναι ηθικό. Άλλο θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε μεγάλε πολυεθνικές που θεωρούν ότι είναι πάνω από τον νόμο, πάνω από τα κοινοβούλια. Το, η McDonald's είναι ένα παράδειγμα. Δεν πληρώνει φόρο στην Ευρώπη. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Nike χρησιμοποιεί θηγατρικέ που βρίσκονται σε ε, κάποιε χώρε ε, σε χώρες ε, offshore, τόσο ώστε να πληρώνει λίγο φόρο. Δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το πόσο δημιουργικές είναι αυτές τις πόσο εφάνταστες είναι, ούτως ώστε να παρακάνουν τον νόμο για να κερδίσουν. Παρακάμπτουν και τις ρυθμιστικές ε, αρχές. Είναι τεράστια φοροδιαφυγή. Αυτό που θα να ξέρω είναι οι επιχειρήσεις πώς βλέπουν την αποτελεσματικότητα των σχετικών νόμων. Πάνω σε αυτό σας ρωτώ, πώς νομίζετε ότι θα σας επηρεάσει αυτή η ευρωπαϊκή πρόταση για το BEPS όσον αφορά δηλαδή τον εταιρικό φόρο την κοινή βάση ε, το εμπόριο, το πηγαίνουμε κρασμόντα, επίση πώ βλέπετε το θέμα του ελέγχου των ξένων εταιρεών. Τώρα, ιδίω μια ερώτηση για την κυρία Τζόνσον. Αποφάσισε η ΝΑΚ να πάει στι ε, κάτω χώρε. Αυτό έγινε ε, λόγω του, του, του φιλικού φορολογικού περιβάλλοντος στη χώρα αυτή. Και είπατε ότι τελικά ακούσατε τη φωνή των καταναλωτών σα, των πελατών σας. Τι σημαίνει αυτό για σας, ότι οι καταναλωτέ συμφωνούν με τέτοιες ε, πρακτικές, ούτω ώστε να μπορείτε να φοροδιαφύγετε κατά δισεκατομμύρια. I would like to clarify something that may... Κυρία Γκέιτ, κοιτάξτε, νομίζω ότι υπήρξε κάποια παρερμηνία ε, στην ερώτησή σας εμεί καταβάλουμε τον φόρο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όπου αναπτύσσουμε δραστηριότητα. Αυτά τα τρία δις που πλώσαμε ως εταιρικό φόρο την τελευταία πέντα αιτία αντικατοπτρίζουν τους φόρους που αντιστοιχούν στα κέρδη των εστιατορίων μας που λειτουργούν σε όλες τις χώρες. δεν θεωρώ, δεν περιμένω κάποια σημαντική στροφή στην ε, πολιτική μας σε σχέση με τη φορολογία σαν αποτέλεσμα ε, αυτών των νέων ευρωπαϊκών νομοθετημάτων κατά της προδιαφυγής ή οτιδήποτε άλλο συναφούς μέτρο. Ε, γιατί εμείς όπως και σήμερα και στο μέλλον θα καταβάλουμε τους φόρους μας αναλογούν. Όσον αφορά τώρα το CCTV, αυτή τον εταιρικό φόρο και κοινή βάση, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά όπως προανέφερα, ο στόχος είναι απλούστευση και διαφάνεια. Εμείς αυτά πρεσβεύουμε. Πάντως, όσον αφορά τις λεπτομέρειες του συστήματος, θα πρέπει να δούμε σε ποια επιχειρηματικά μοντέλα θα αντιστοιχεί αυτή η ρύθμιση, να τα καλύπτει όλα και να υπάρχει ισότητα. Τώρα, όσον αφορά ε, την επιδίωξη της διαφάνειας αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει. Τζόνσον, για την Nike. Ευχαριστώ για την ερώτηση για τους ε, καταναλωτές μας. Παρακολουθούμε συνεχώς τις προτιμήσεις των καταναλωτών και την συμπεριφορά τους απέναντι στην εταιρεία μας. Αυτό αλλάζει ε, μέρα με τη μέρα και ανάλογα με το θέμα. Mm. Οπότε δεν μετράμε τις ε, προτιμήσεις τους σε σχέση με τη φορολογία μας ή οτιδήποτε άλλο αφορά τα Paradise Papers. Όσον αφορά την ε, νομοθετική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ένα αποτελέσματα, εμείς είμαστε υπέρ ε, φορολογικής μεταρρύθμισης που απλοποιεί τις διοικητικές διαδικασίες και καθιστά τον νόμο σαφή. Και είμαστε υπέρ οποιασδήποτε τέτοια κίνηση στην Ευρώπη για την ερώτηση για την Ολλανδία και το πώς συνεργαζόμαστε με την Ολλανδία. Ως ε, χονδρική και λιανική πώληση και ως ε, καινοτόμος εταιρεία ε, ακολουθούμε τις κατευθυντήριες γραμμές του ΩΣΑ που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες για να υπάρχει το κατάλληλο ποσό αμοιβή σε κάθε χώρα σύμφωνα με τις υπηρεσίες και το τι επιτυγχάνει και η εταιρεία αυτή στην κάθε χώρα. Ε, δεν μου απαντήσατε για τους υπαλλήλους σας ε, στις Βερμούδες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πλέον εταιρείε στην ε, Βερμούδα. Είμαστε στην διαδικασία κλεισίματος των εταιρείων αυτών. Μάλιστα, η FTD, David Coburn. Μάλιστα. Ακούγοντας αυτήν την ε, επιτροπή εδώ πέρα των ε, Ροβεσπιέρων, δεν μου προξενεί έκπληξη που το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να μετακινηθεί στην Βρετανία. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Και είμαι σίγουρος ότι μετά το Brexit θα δείτε και άλλες εταιρείε να μετακινούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καλό αυτό για μας. Οπότε το Brexit θα είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν τους αδικό. Υπάρχουν καλοί λόγοι να έρθει κανεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα τα ξέρουν αυτά οι κυρίε. Ο φόρο ε, και βεβαίω και το νομικό σύστημα είναι καλύτερο. Γι' αυτό οι περισσότερε εταιρείε στον κόσμο, όταν κάνουν κάποιε εταιρείε, ε, θέλουν ε, να ισχύει το βρετανικό δίκαιο. υπάρχει ένα απλό λόγο. Είναι σαφέ και δεν είναι προκατηλημένο και λειτουργεί. Και όπω είπε και η κυρία, και η γλώσσα παίζει ρόλο. Και το ίδιο ισχύει και στο Delaware. Γι' αυτό κάνουν και εκεί εταιρείε. Ε, και υπάρχει ένα απλό λόγο όμω. Οι περισσότεροι εδώ μέσα δεν έχουν εργαστεί ποτέ σε εταιρεία και δεν έχουν διευθύνει ποτέ του εταιρεία και δεν έχουν ιδέα. Οπότε οι επιχειρήσει δεν υπάρχουν για να πληρώνουν φόρο. Οι επιχειρήσει δημιουργούνται για να έχουν κέρδη και απασχολούν και κόσμο επευκαιρία. Και οι δύο εταιρείε αυτέ μπορεί να έχουν περιπλοκέ δομέ, αλλά τουλάχιστον απασχολούν πολλού ανθρώπου στην Ευρώπη κάτι το οποίο δεν κάνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείε ή η Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολείται με το να καταστρέφει θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Και πραγματικά ελπίζω να φέρετε περισσότερες επιχειρήσεις στην Βρετανία. Ευχαριστώ. Η ερώτηση λοιπόν είναι θα φέρετε περισσότερες επιχειρήσεις και έργο στην Βρετανία. εντάξει και οι άνθρωποι δεν υπάρχουν μόνο για να πληρώνουν φόρους, αλλά το πληρώνουν. Όχι, κοιτάξτε, οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρώνουν ελάχιστο φόρο. Είναι, αυτό είναι φορολογικό καθεστώς. Το καλύτερο ίσως. Όχι, πληρώνουν λιγότερο από τους υπόλοιπους πολίτες. η McDonald's έχει έναν ε, θελημένο στόχο να βγάζει κέρδη και βεβαίω και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όσον αφορά την Nike, ελπίζουμε και εμείς να αναπτυχθεί η εταιρεία μας στο Ηνωμένο Βασίλειο και να προτιμούν ε, οι καταναλωτές τα προϊόν μας. Ωραιότατα. Από το ΕΛΚ, Ντάριος Ροζάτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τις δύο κυρίες που ήρθαν σήμερα εδώ. Και εγώ βεβαίω είμαι καταναλωτής ε, των McDonald's, έχω και τρία ζευγάρια Nike στο σπίτι και ελπίζω και στο μέλλον να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσω με σας κυρία Γκέιτς. Είπατε ότι η McDonald's πληρώνει φόρο σε κάθε κράτο μέλος όπου λειτουργεί. Δηλαδή σε όλα τα κράτη μέλη. Η ερώτηση μου είναι η εξή: Το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρεία σας βασίζεται σε ένα μοντέλο δίκαιο ε, και σας πληρώνει πνευματικά δικαιώματα ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου σε ποιον, στο, στην έδρα του Ηνωμένου Βασιλείου πρώην ε, Λουξεμβούργου. Πρώτη ερώτηση είναι αυτή και δεύτερη. Πόσο κέρδος του απομένει αφού πληρώσει αυτά τα πνευματικά δικαιώματα. Ποιο είναι το ποσοστό δηλαδή των πληρωμών αυτών ε, σε κάθε χώρα που ε, δραστηριοποιούνται τα μοτινότητα. Δηλαδή πόσο από αυτό το κέρδος παραμένει στις χώρες. Και μετά αντιλαμβάνομαι ότι πληρώνεται φόρους σε αυτό το υπόλοιπο. Πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Δεύτερη ερώτηση έχετε κάποια συγκεκριμένη συμφωνία φορολογική με κάποιο κράτος μέλος ε, της Ένωσης. Είχατε τέτοια συμφωνία με το Λουξεμβούργο. Έχετε τέτοια συμφωνία με το Ερμένο Βασίλειο ή με άλλο κράτος μέλος. Και προς την ε, κυρία Τζόνσον, εάν μου επιτρέπετε, έχουμε, έχω μία παρόμοια ερώτηση. Ποιο είναι το ποσοστό των ε, πνευματικών δικαιωμάτων, ακριβώς, σε σχέση με τον συνολικό τζίρο και με το, τα κέρδη προφόρων. Και η άλλη ερώτηση είναι ποιο είναι ο πραγματικός συντελεστής ε, φόρου στο κέρδος ε, στην Ευρώπη και τέλος είπατε ότι πληρώσατε φόρους τις είπα, σε όλα τα επαναπατρισμένα κέρδη, εάν κατάλαβα καλά. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό ότι όλα τα κέρδη που έχουν μεταφερθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τελικά φορολογήθηκαν ε, στη ΣΥΠΑ ή όχι. Ναι, κυρία Γκέιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τα πνευματικά δικαιώματα που, και τα δικαιώματα δικαιώσεις που πληρώνουν οι εταιρείε McDonald's και χρήστε του σήματο πληρώνονται είτε στη ΣΥΠΑ είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο παγκοσμίω. Και όταν μιλάω για τα κέρδη που παραμένουν στην McDonald's, μιλάμε για 15% του τζίρου μόνο, γιατί έχουμε, όπως σας είπα, 85% με franchise. Και πληρώνουν επίσης ε, φόρους ε, οι κάτοχοι των ε, εστιατορίων στις χώρες τους. Δεν έχω ακριβή νούμερα για την Ευρώπη, αλλά 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 5 χρόνια είναι μέσο όρο 29% ως συντελεστής και όπως ξέρετε διαφέρουν πάρα πολύ οι συντελεστές από χώρα σε χώρα. Όσον αφορά τώρα μεμονωμένες ε, συμφωνίες, ε, μπορώ να επαναλάβω ότι δεν έχουμε συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο, φορολογικές για το θέμα του Λουξεμβούργου είναι ένα θέμα το οποίο ερευνάται αυτήν την ε, στιγμή και και θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπατε, δεν μπορώ να το συζητήσω. Να απαντήσω στην τελευταία σας ερώτηση, η πρώτη. Ο νέος φορολογικός νόμος της ΕΠΑ απαιτούσε να πληρώσουμε φόρο τον λέμε μεταβατικό φόρο, άλλοι το λένε διόδια, να πληρώνουμε φόρους στα μη επαναπατρισμένα κέρδη οπουδήποτε ανά την Οπότε έχουμε κέρδη σε ένα κράτος ε, τα οποία δεν έχουν επαναπατριστεί στις Είπα υπόκεινται σε φόρο. Είναι περίπλοκος ο υπολογισμός, αλλά η βάση του υπολογισμού είναι το ότι τα κέρδη αυτά στο εξωτερικό. Δηλαδή και επανεπενδύσεις που έγιναν, παραδείγματος χάρη, στο κέντρο διανομής του Βελγίου. Και αυτά έχουν φορολογηθεί πλέον στις ΗΠΑ επειδή δεν επαναπατρίστηκαν. Στα γραπτά μου σχόλια επίσης ε, λάβαμε την ερώτηση για το ποσοστό των πνευματικών δικαιωμάτων ως ποσοστό του τζίρου και είπα ότι δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο παρακολουθούμε ή αποκαλύπτουμε. Έχουμε εξωτερικά πνευματικά δικαιώματα, τρίτα μέρη και εσωτερικά, αλλά δεν τα παρακολουθούμε. Το, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής στην Ευρώπη δεν το παρακολουθούμε, μπορούμε να το υπολογίσουμε και να σας το δώσω μετά. Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ κυρίε σε σχέση με την τελευταία απάντηση που δώσατε, αν αγοράζω παπούτσια στις Βρυξέλλες, τι ποσοστό αποδίδει στην αρχή πνευματική ιδιοκτησία η Ναϊκή. Πάει στο Όρεγκον ή στι Βρυξέλλες. Στο Όρεγκον πάει. Κατά μέσο όρο, τι ποσό αφορά την πνευματική διοκτησία για τα προϊόντα της ΝΑΚΙ. Δεύτερη ερώτηση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια μαύρη λίστα και μια γκρι λίστα για τους φορολογικούς παραδείσους. Οι εταιρείε σας έχουν φυγατρικές υποκαταστήματα σε εκείνες τις χώρες. Τρίτη ερώτηση τι ποσοστό από το σύνολο των φόρων που καταβάλουν οι εταιρείε σας έχουν καταβληθεί στις Βερμούδες. Ποιο είναι το ποσοστό από το συνολικό φόρο που έχει καταβάλει, έχει πάει στις Βερμούδες. Επίσης, σε κάθε φορολογική αρχή, κάθε χώρα της Ένωσης, σε σχέση με τις εκθέσεις αναχώρα. Υποβάλλεται σε αυτές τις φορολογικές ε, αρχές το τι ισχύει όσον αφορά ε, το τι φόρο καταβάλλεται. Αυτές είναι οι ερωτήσει μου, Πρόεδρε. Κυρία Τζόνσον, έχετε το λόγο. Σε σχέση με την ερώτησή σας για την αναχώρα έκθεση, να απαντήσω αυτό το υποβάλλουμε όσον αφορά το τι φοροκαταβάλλουμε στην κυβέρνηση των ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Ακριβώς όπως επιβάλλει το Αμερικανικό Δίκαιο. Τώρα για Βρυξέλλες. I'm going Τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Θα στα τα πω αναλυτικά γιατί έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις στις Βρυξέλλες. Στο Βέλγιο, ενώ. Έχουμε μια επιχείρηση για την ε, διανομή που καλύπτει όλο τον κόσμο και αυτός ο διανομέας πληρώνει αυτά τα οποία πρέπει να πληρώνει μια τέτοια εταιρεία. Και επίσης αυτό αντικαθευδίζεται και στο τι πρέπει να μα δίνουν οι τρίτοι που κάνουν αυτή τη δουλειά. Τώρα όσον αφορά ε, ένα ζευγάρι που πουλάει κάποιο χονδρέμπορο σε κάποιον λιανέμπορο στι Βρυξέλλε. ή τι πληρώνουμε σε κάποιον τρίτο. Έχουμε 500 στο Ηνωμένο Βασίλειο και τελικά οι λιανοπολιτές μας για τα παπούτσια θα χρειώσουν το ίδιο στις Βρυξέλλες όπως και εάν πουληθούν τα βούσια μας από κάποιο κατάστημα που δεν είναι της ΝΑΕΚΕ. Τώρα για το τι ποσοστό των φόρων μας έχει πληρωθεί στις Βερμούδες. Ε, υπάρχει μία επιβάρυνση 2 εκατομμύρια και πληρώθηκε ο φόρος της αλλαγής του μετασχηματισμού εκεί. Yates. Συμφωνώ με τόσο είπε η Νάγκη όσον αφορά τις εκθέσεις γιατί και εμείς αυτό κάνουμε στις ΗΠΑ όσον αφορά την εκεί εφορία για το τι καταβάλουμε. Για το 17. Επίσης, επιχειρούμε σε 120 χώρες με ναι. τους συμβασιούς δικαιόχρησης ή όχι. Και έχουμε, όπως είπατε, κάποιες εταιρείες που βρίσκονται στις χώρες της γκρίζας λίστας. Αλλά θα ήθελα να με ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο παράδειγμα χώρα για να σας απαντήσω. Τώρα όσον αφορά τις Βερμούδες. Εκεί καταβάλλεται ο φόρος για τις εμπορικές δραστηριότητε που λαμβάνουν εκεί χώρα και επίσης έχουμε εκεί και κάποια ασφαλιστική εταιρεία και αυτή φορολογείται εκεί. Επιρώτηση του κύριου Χαροκή. Εάν κατάλαβα καλά για την αναχώρα έκθεση, τελικά αυτή την έκθεση την υποβάλλεται όχι στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές χώρες, μόνο στη ΣΥΠΑ. Έτσι, καλά κατάλαβα. Δεν υποβάλλεται τέτοιου έκθεση, τέτοιες πληροφορίες ανά χώρα στην Ευρώπη. Μόνο στη ΣΥΠΑ. Σύμφωνα με τους κανόνες του ΟΣΑ και την πολιτική που έχουμε για τη φορολογία ανταλλάσσουν τις πληροφορίες οι φορολογικές αρχές των ευρωπαϊκών χωρών. και όποια ευρωπαϊκή χώρα θέλει παραπάνω πληροφορίε μπορεί να απευθυνθεί στι φορολογικέ αρχέ των ΗΠΑ. Ναι, ναι, δεν έχω προσθέσει τίποτα, λέει η κυρία Χέιτ. Και τώρα. Έχουμε ώρα για το κατσιδιά. Έτσι μπορούμε να επανέλθουμε με κάποιες ερωτήσεις που θεωρήσατε ότι αν και υπευλήθησαν δεν καλυφθήκατε. Ο συνεισηγητής, ο κ. έχετε το λόγο. Uh, let me Να επανέλθω στην πρώτη μου ερώτηση γιατί απογοητεύτηκα λίγο διότι δεν άκουσα απάντηση ή η απάντηση είναι διαφορετική από αυτή που ε, θα άξιζε στην ερώτησή μου. Λόγω νομοθετικών και μη νομοθετικών αλλαγών στην φορολογική επικράτεια, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά παγκοσμίω, εταιρείε όπω οι δικέ σας επανεξετάζετε την προσέγγιση σας στην φορολογική πολιτική. Δεν ε, λέω ότι δεν είχατε ποτέ τη λογική ότι η business ακολουθεί τον φόρο, αλλά και ανάποδα να είναι υπάρχουν διάφορες επιλογές ό,τι αφορά την προσέγγιση στο φορολογικό θέμα. Εδώ έχω την αίσθηση ότι η εγκατάλειψη της Βερμούδας από την εταιρεία σας είναι λόγω της ε, αλλαγής στη φορολογική νομοθεσία των ΗΠΑ. Και για σας η δραστηριοποίηση στο Λουξεμβούργο δεν ήταν λόγω φορολογικών ρυθμίσεων που σας εκχώρησε, μάλλον ήταν λόγω φορολογικών ε, εκχωρήσεων που σας έκανε η ε, λουξεμβουργική κυβέρνηση. Είναι σημαντικό για τους συναδέλφους μου και εμένα να γνωρίζουμε αν έχετε επανεξετάσει το θέμα αυτό και αν επιδιώκετε τώρα περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη σαφήνεια σε φορολογικά θέματα και προσπαθείτε να συμμορφωθείτε με την αρχή ότι θα πρέπει να πληρώνετε φόρους και σε κάποιε από τους τόπου που ε, δραστηριοποιήσετε και δεν μιλώ για φόρους για την έγκυο περιουσία την οποία διατηρείτε στις χώρες αυτές, αλλά ε, για ε, φόρους επί των κερδών που αποκομίζεται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις συγκεκριμένε χώρες. Η εκπρόσωπος της ΝΑΕΚΕ Σύμφωνα με τι κατευθύνες γραμμέ του ΩΣΑ, υποχρεώμεθα να καταβάλουμε φόρο σύμφωνα με την αξία που δημιουργείται σε κάθε δικαιοδοσία όπου δραστηριοποιούμεθα επιχειρηματικά. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε έσοδα σε μία δικαιοδοσία ε, χωρίς ε, να παραπονηθεί κάποια άλλη δικαιοδοσία ότι έχασε έσοδα. Ακολουθούμε λοιπόν την αρχή αυτή, αναγνώριση ε, των κερδών εκεί όπου δημιουργείται η αξία η συνολική μας φορολογική επιβάρυνση περιλαμβάνει και τέλη, κάτι που είναι διαφορετικό από την υπόθεση του McDonald's. Θα ήθελα να αντιληφθεί η Επιτροπή σας ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για μια επιχείρηση όπως η ΝΑΕΚΕ. Και ως τώρα αυτό δεν συζητήθηκε στην παρούσα συζήτηση. Κύριε. όπως πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, αναθεωρούμε διαρκώς την εταιρική μας δομή στην βάση φορολογικών και άλλων ρυθμίσεων για να διατηρήσουμε αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα. Συνεισηγητής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση ακόμη, ο κ. Κοφούτ. Κύριε Γέιτς, ρώτησα για τις δομές σας. Δεν απαντήσατε καθαρά. Μπορείτε να απαντήσετε καθαρά με ναι ή όχι. Η νέα περίπλοκη δομή που έχετε δημιουργήσει έχει σχέση και με φορολογικά θέματα, ναι ή όχι. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, δευτερο οταν ρωτώ για τις κινήσεις κλπ. Εσείς η ίδια αναφερθήκατε στην, ε, αν, στην έκθεση Unhappy Meal. Εσείς άλλωστε μιλήσατε πρώτοι για αυτήν. Θα ήταν ε, σημαντικό και για την Επιτροπή μας και για το Κοινοβουλίο να έχουμε μια γραπτή απάντηση εκ μέρους σας. Εκ μέρους σας. Δηλαδή, ποιες ανακρίβειες έχετε εντοπίσει στην έκθεση αυτή για να μπορέσουμε να τη συζητήσουμε. Εάν λέτε ότι υπάρχουν ανακρίβειες, νομίζω μπορείτε να τοποθετηθείτε και γραπτός. Εάν όχι, τότε δεν κατανοώ το σχόλιο σας. Και τέλος, και για τις δύο κυρίες, είστε εσείς και οι επιχειρήσεις σας υπέρ περισσότερης διαφάνειας στα φορολογικά θέματα. Για παράδειγμα, δημοσιοποίηση των εκθέσεων αναχώρα για κάποια βασικά νούμερα, ώστε να είναι διαφανέστερο για το κοινό, να αντιληφθεί το κοινό δηλαδή πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις σας. Ε, ε, θα, θα, μπορούσατε να υποστηρίξετε λοιπόν ε, αυτή την διαφάνεια στις εκθέσεις αναχώρα. Η κυρία Γίτς. Η τρέχουσα δομή της McDonald's στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει δημιουργηθεί και πληρώνει τους φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο για ο κάθε είδου εισόδημα που αποκτά εκεί. Δεν έχει καμιά σχέση με οποιασδήποτε ειδικέ φορολογικέ αποφάσει. Σε ό,τι αφορά, tax rulings δηλαδή, ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση των εκθέσεων αναχώρα, η δική μας προτίμηση είναι η έκθεση αυτή ε, να μπορεί να διαβιβάζεται μεταξύ φορολογικών αρχών, διότι υπάρχουν και ευαίσθητα στοιχεία μέσα σε αυτές τις εκθέσεις για την McDonald's. Λειτουργούμε σε πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν πάνω από 950.000 εστιατόρια ταχυφαγίας σε όλη την Ευρώπη σήμερα μικρές επιχειρήσεις που δεν ε, έχουν ωστόσο να αντιμετωπίσουν τις ίδιες απαιτήσεις όπως η McDonald's λόγω της νομοθεσίας. Αναμένουμε ότι η έκθεση Unhappy Meal σε ό,τι αφορά αυτήν θεωρώ ότι απάντησα στις ουσιώδεις ερωτήσεις και πάλι δεν είμαι βεβαία ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερα θετικό στοιχείο αν καθίσω να την ε, διεξέλθω γραμμή προς γραμμή για να σας δώσω ε, συγκεκριμένα στοιχεία. Ως επιχείρηση πληρώνουμε τους φόρους μας. Δημιουργούμε απασχόληση, προσλαμβάνουμε κόσμο, επενδύουμε. Πιο σημαντικό για μένα είναι να περάσει το μήνυμα της McDonald's προς τα έξω και να εξηγήσει τι κάνουμε αντί να αρχίσουμε να ας πούμε, ασχολούμεθα με άλλα θέματα. Ο κ δεν αντιλαμβάνομαι γιατί αυτή η μυστικότητα. Γιατί τηρείται μυστικότητα γύρω από τις ε, ανακρίβειες που έχετε, που έχετε εντοπίσει στην έκθεση δυστυχές γεύμα. Ε, θα μπορούσε το κοινό να πληροφορηθεί. Δεν θα έπρεπε να ξεχαριστεί. Θα λάβω υπόψη μου το αίτημά σας, απαντάει η κυρία Γέιτς. Η κυρία Τζόνσον. Έχουμε καταθέσει τώρα την πρώτη μας έκθεση αναχώρα. Στην παρούσα φάση, ο τρόπος με τον οποίο συντάσσεται η έκθεση, θεωρώ ότι δεν είναι κατάλληλη έκθεση για ε, υποβολή στο κοινό. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει η φορολογική αρχή την έκθεση αναχώρα. Και θα πρέπει να δούμε αν όλες οι χώρες σέβονται και, και θα δούμε λοιπόν πώς θα, πώς θα ε, λάβουν υπόψη τις εκθέσεις αυτές οι φορολογικές αρχές. Για την ώρα πληρώνουμε φόρους σε όλες τις δικαιοδοσίες όπου δραστηριοποιούμεθα παγκοσμίω. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Ευχαριστώ προσκεκλημένες μας. Με βάση την ε, σημερινή συζήτηση μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και οι πληρών πληρώνουν φόρους. Όμως δεν είναι σαφές εάν πληρώνουν αναλογικά το ίδιο με τους μικρότερους ανταγωνιστές τους που είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην ίδια αγορά θα ήθελα να ρωτήσω και τις δύο κυρίες εάν ε, χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα σε διάφορες ε, χώρες ή εάν ε, συμμετέχουν σε προεκλογικές εκστρατείες και αν ναι σε ποιες χώρες και με ποια ποσά. Η κυρία, Γε, η κυρία Τζόνσον. Με συγχωρείτε, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά ευχαρίστω να σας απαντήσω αργότερα. Το ίδιο κι εγώ. Ναι, είναι βεβαίως και εκτός ε, του αντικειμένου της Επιτροπής μας. Τέλος πάντων, Πίτερ Σίμων. Η ερώτηση μου προς την κυρία Γέιτς. Κυρία Γέιτς, ε, είπατε και στις γραπτές σας απαντήσεις ότι μεταξύ 2013 και 2017 πληρώστε πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια, είπα, ε, φόρο επιχειρήσεων, ένα μέσο όρο 29% δηλαδή. Μπορείτε να μας το εκτιμήσετε κάπως καλύτερα αυτό, να μας πείτε δηλαδή με αριθμούς ε, πώς ήταν η φορολογία της επιχείρησής σας πριν από την αναδιάρθρωση και πόσοι μετά και μπορείτε να μας δώσετε μια γενική εικόνα για το πόσους φόρους πληρώνατε πριν και μετά με βάση ποιο κέρδος και ποιο τζίρο. Κυρία Γέιτς. Σε μία από τις προηγούμενες ε, απαντήσεις μου είχα πει πως ε, το νόμο ποσοστό για την πενταετία στην McDonald's ήταν 27% οπότε αυξάνεται τώρα ο συντελεστής όμως αυτό οφείλεται και στην ε, ανάπτυξη της εταιρεία. Δηλαδή αν το σκεφτείτε αν μια εταιρεία με υψηλότερο συντελεστή αναπτύσσεται περισσότερο από μια χώρα με χαμηλότερο συντελεστή αυξάνει και το μέσο όρο μας αυτό. Υπάρχει και επιπρόσθετος φόρος που πληρώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της μετακίνησης ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί κάποια πνευματική ιδιοκτησία που βρισκόταν ε, στην Ασία μετακινήθηκε τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε έχουν αυξηθεί και οι φόροι που πληρώνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κ. Σίμων θέλει να επανέλθει έχετε έτοιμους τους αριθμούς ή μπορείτε να μας στείλετε μετά πόσο φόρο πληρώσατε σε σχέση με ποιο κέρδος και ποιο τζίρο. Αυτά τα στοιχεία. Ε, δεν τα έχω πρόχειρα. Τα παρακολουθούμε ως σύνολο. Ο τζίρος που περιλαμβάνεται και είναι δημοσιεύσιμος είναι ανακλάδο και όχι γεωγραφικά γιατί αλλάξαμε όπως σας είπα επιχειρηματικό μοντέλο δεν έχετε αυτές τις πληροφορίες αυτή τη στιγμή ή μπορείτε να μας ε, τις στείλετε μετά έχουμε υποχρέωση και υποβάλλουμε οτιδήποτε απαιτεί ο νόμος. Αλλά αναχώρα τον τζίρο και τα έσοδα δεν ε, είναι κάτι το οποίο κανονικά δημοσιεύουμε, είναι εμπιστευτικό. Μάλιστα, σαφές. Η κυρία Τζόνσον, θέλετε να απαντήσετε. Δεν θυμήθηκε κάτι σε μένα. Ωραία. Μαντάριος Ροζάτη. Κυρία Γέιτς, να επανέλθω στην προηγούμενη ερώτησή μου. Είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είπατε ότι οι κάτοχοι της δικαιόψης ε, πληρώνουν 85%. Τι εννοείτε, ε, αυτό είναι το κέρδος, τίνος πράγματος δηλαδή, του κέρδους. Και σημαίνει ότι μιλήσετε για μία μέση φορολογία 29% στην Ευρώπη. Αυτό είναι 29% του 15% που απομένει. Ναι, ναι, να το ξεκαθαρίσω, γιατί δεν εννοούσα αυτό. Σήμερα η McDonald's. Δηλαδή, αν σκεφτείτε τον αριθμό των εστιατορίων, 15% των εστιατορίων είναι η ιδιοκτησία τη εταιρεία, 85% είναι η ιδιοκτησία ιδιωτών, που είναι ανεξάρτητοι επιχειρηματίες, έχουν μια επιχειρηματική ελευθερία. Βεβαίω πάντα εντό τη ε, νομοθεσία. Δεν έχω πληροφορία για τα τρίτα μέρη, για τα φορολογικά τους. Ναι. Αυτά τα τρίτα μέρη που είπατε. Ναι, ναι, είναι ανεξάρτητοι επιχειρηματίες. Αλλά έχετε συμφωνίες μαζί τους. Βάση των οποίων λειτουργούν ε, τα, τα εστιατόρια με το σήμα σας. Ναι, και πληρώνουν γι' αυτό. Σωστά. Ε, πόσο πληρώνουν. Ε, Διαφέρεων αυτά. είπαμε το πώς συλλέγονται τα πνευματικά δικαιώματα. Το, αν το ερώτημά σας είναι το εάν έχουμε πληροφορίες για τους φόρους που πληρώνουν αυτοί, δεν τους έχουμε. Η συμφωνία απαιτεί να τηρούν ε, τα νόμιμα και τη φορολογική νομοθεσία. Ναι, ναι, για το 29% ε, ποσοστό φόρο. Αυτό ισχύει για την δική μας τη λειτουργία και για φόρο επί των πνευματικών δικαιωμάτων που λαμβάνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ένα συνολικό ευρωπαϊκό νούμερο. Δεν έχετε δηλαδή μια ιδέα του τι ποσοστό του κέρδους προφόρων ε, είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Γιατί μειώνουν την φορολογική βάση στα κράτη-μέλη. Ε, αυτή την πληροφορία θα ήθελα. Η πληροφορία την οποία μπορώ να σας ε, δώσω όσον αφορά τις πληρωμές από τα τρίτα μέρη σε σχέση με την εταιρεία είναι ότι η McDonald's το 2017, το 2017 είχε έσοδα 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχεδόν και παγκοσμίω έχουμε 12 δισεκατομμύρια πωλήσει της εταιρεία και πάνω από 10 δις ε, πληρωμές ε, ε, πνευματικών δικαιωμάτων από τους συμβαλόμενους. Αυτό το οποίο πρέπει να αντιληφθείτε για το franchising είναι ότι η πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων τους δίνει τη δυνατότητα να τυχθούν γρήγορα και επικερδώς. Αν σκεφτείτε τις 425.000 άτομα που απασχολούνται, απασχολούνται και από την McDonald's και τα ανεξάρτητα εστιατόρια και τους εστιατόρες. Πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα για να λάβουν το σήμα, την τεχνογνωσία, την καινοτομία και την πρόσβαση σε πολλά ωφέλη που δεν χρειάζεται να δημιουργήσουν μόνοι τους και αυτό κατά κανόνα σημαίνει υψηλότερα κέρδη από το να ξεκινούσαν μια επιχείρηση μόνοι τους και να δούλευαν χωρίς το σύστημα των McDonald's και τα 60 χρόνια επιτυχίας που σημαίνει αυτό. Κυρία Παλώμα Λόπες Μπερμέχο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγκεκριμένη ερώτηση που την υπέβαλα αλλά δεν απαντήθηκε. Να την επαναδιατυπώσω αν δεν έγινε κατανοητή. Πώς θα επηρεάσουν οι νομοθετικές αλλαγές όσον αφορά την πληρωμή των φόρων σε αυτές τις δύο ε, εταιρείε όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, πώς θα επηρεαστούν και πώς θα διαρθρωθεί αυτή η νέα κατάσταση. Τι έχετε προβλέψει η εταιρεία σας σε σχέση με αυτές τις α, άλλαγες όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγγνώμη, αλλά δεν κατάλαβα αυτές τις νομοθετικές αλλαγές σε σχέση με τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας. Μήπως εννοείται τις νομοθετικές αλλαγές στα δικαιώματα, στα ψηφιακά. Γίνεται πολύ κουβέντα, αλλά δεν έχω καταλάβει τι μας ρωτάτε. Ούτε εγώ, λέει η, κυρία από την Μακδόναλτ. About, about, ε, Μήπως λέτε για εσωτερικές ε, αλλαγές ε, στην εταιρεία Μπρίμεχο. Επιμένω να σας το πω με άλλα λόγια. Το Κοινοβούλιο ε, έχει αυτή την κοινή βάση όσον αφορά τι εταιρείες και τη φορολόγηση και όσον αφορά τον έλεγχο των ξένων εταιρείων. Θέλω να καταλάβω ακριβώς πως η αλλαγή που θα γίνει τώρα, η νομοθετική, πρόκειται να επηρεάσει τα δικαιώματα που καταβάλλονται στις εταιρείες σας. Johnson, ναι, πληρώνουμε σε κάθε χώρα που προβλέπει η νομοθεσία της και ανάλογα με το τι προβλέπει ο ΣΑ. Δεν νομίζω να υπάρξει κάποια αλλαγή για την φορολόγησή μας, για το τι καταβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά λειτουργούμε σε όλες τις χώρες και όπου λειτουργούμε πληρώνουμε φόρους. Δεν θα αλλάξει τίποτα με τους νέους κανόνες. Well, other... έχουμε άλλες ερωτήσεις. Όχι. Οπότε, τώρα πεθαίνουμε στους συνεισηγητές. Αν έχουν κάποιες παρατηρήσεις... Κύριε Κόφοντ, απλώς να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στην Επιτροπή μας και ελπίζουμε να συνεχιστεί η συνεργασία μας όσον αφορά να φωτίσουμε τα πράγματα. Δυστυχώς δεν ισχύει αυτό με όλους όσους προσκαλούμε. Ελπίζω να έχει συνέχεια η επαφή μας για αυτά τα θέματα. Βεβαίως, βεβαίως λέει η κυρία Γιέτς. Τώρα οι προσκεκλημένες μας μήπως θέλουν να προβούν σε κάποια καταληκτική παρατηρήση επί τη βάση των όσων συζητήσαμε. Έχετε κάποια δήλωση που θέλετε να κάνετε. Δεν είναι υποχρεωτικό. Γιέτς. Ναι, ναι, ναι, έχω μια σύντομη δήλωση. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δώσατε για την πρόσκλησή σας προς την ε, McDonald's. Εμεί αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρχει μια συνεχιζόμενη συνεργασία που να διακρίνεται από διαφάνεια που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, μα πρόβλημα σε κάποια δήλωση όσον αφορά τις ε, εξελίξει στην πολιτική, γιατί θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει προς απλούστευση στην νομοθεσία, προ διαφάνεια. Ε, για όλα τα φορολογικά θέματα επίσης θεωρούμε ότι είναι πολύτιμα σε αυτές οι αρχές, σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειες που καταβάλλατε σχετικά. Και εσείς, κυρία Τζόνσον, και εγώ και εγώ συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Αγία και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε να έρθουμε σήμερα εδώ ή να εκεί. Αυτό το οποίο πρεσβεύει είναι μια φορολογική πολιτική που θα βοηθά το επιχειρηματικό κλίμα, θα διέπεται από απλούστευση, συνέπεια, και που αυτό θα ισχύει σε παγκόσμια κλίμακα. Να ισχύει η φορολογική πολιτική παγκόσμια. Αυτό θέλουμε. Και γι' αυτό και θέλουμε να συμβάλλουμε στην προβληματική. Ο πρόεδρος. Δεν θέλω να πιστεύω στις λεπτομέρειες όσο συμπεράσματα γιατί νομίζω όλοι θα κάτσουμε να σκεφτούμε όλα αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα. Και όλα όσα ακούσαμε θα τα αποτυπώσουμε στο τελικό κείμενο της Επιτροπής. Πολλά ακόμα θα πρέπει να διερευνήσουμε, πολλά θα πρέπει να γίνουν ε, ακόμα και από πλευράς ε, ερευνητικής δημοσιογραφίας. Πάλι ανέκυψαν ε, αποκαλύψεις, αλλά και εμείς οι νομοθέτες θα πρέπει να δουλέψουμε, θα πρέπει να θωρακίσουμε το νόμο Ευχαριστούμε και την κυρία Τζόνσον και την κυρία Γιέτς που ήρθαν σήμερα. Και όσον αφορά τις εταιρείε που δεν αποδέχονται την πρόσκλησή μας, αυτό έγινε για διαφορετικούς λόγους όσον αφορά τον καθένα. Αλλά όπως είπα στην ε, αρχή, ε, είπαμε ότι οι συντονιστές των υπόλοιπων ομάδων θα αναζητήσουν λύσεις ούτω ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Και πάλι σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Τώρα, σας ανακοινώνω ότι οι δύο συνεισηγητές μας οργανώνουν μια συζήτηση με μορφή πάνελ για τις μεταρρυθμίσεις Τραμπ στα φορολογικά στις 27 Ιουνίου στις 1 παρατέταρτο στο 6Q1, σε αυτό το κτίριο. Το θέμα εννοείται ότι είναι ενδιαφέρον για την Επιτροπή μας και για άλλους. Επόμενη συνεδρίασή μας. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα 25 και 5η 28 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πέρα στη συνεδριάσεις.